Uh, uh, Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να συζητήσω να καθίσετε. Έχουμε την ακρόαση για τα ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στο σημείο 4 στην ε, ημερήσια διάταξη, αλλά όσο κάθεστε εγώ θα ξεκινήσω με κάποιες ανακοινώσεις. Καταρχήν πρέπει να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται θα εγκρίνουμε και τα πρακτικά της συνεδρίας της Δευτέρης ε, Ιουλίου, της 11ης Ιουνίου, της 11ης Ιανουαρίου και της 7ης Δεκεμβρίου του 2017. Εάν δεν έχουμε αντιρρήσεις, εγκρίνονται και τα πρακτικά και θα ήθελα να προχωρήσω και στις ανακοινώσεις. Ε, καταρχήν για τις γλώσσες δεν έχουμε διερμηνία στα κροατικά, δανικά, ε, λετονικά και γέλικ. Όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν και μετά έχουμε και τις συστάσεις των συντονιστών. Καταρχήν ορισμός των ε, ε, συναδέλφων για τις γνωμοδοτήσεις, η κυρία Μακοβέ για το σχέδιο γνωμοδότησης για την Επιτροπή Κοντ, για τις έρευνες που διεξάγει η Όλαφ, σχετικά με τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τη δέχεστε, οκ, okay. ορίζεται λοιπόν και θα ήθελα να σα υπενθυμίσω πω θα γίνει και ηλεκτρονική ψηφοφορία σήμερα στι 6 το απόγευμα. Επίση θα κάνουμε και μια ψηφοφορία μαζί με την Επιτροπή ΕΚΟΝ στο σημείο 12. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να μετακινηθούμε στην αίθουσά τους που είναι σε αυτό το κτίριο, στον τρίτο όροφο η αίθουσα 50. Σας παρακαλώ μην το ξεχάσετε. Δύο ψηφοφορίες λοιπόν στη Λίμπε και μία από κοινού με την ΕΚΟΝ στην άλλη αίθουσα. Δύο μέλη έχουμε μόνο εδώ. Σίγουρα τα ακούσατε λοιπόν. Συνάδελφοι, τώρα που τελείωσαμε τις ανακοινώσεις μπορώ να περάσω στο σημείο 4. Να καλωσορίσω θερμά όλους τους προσκεκλημένους που έχουμε για το σημείο τούτο. Ξέρετε πως το σημείο 4 είναι η ακρόαση για την μήνυ ακρόαση για τα ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην Ευρώπη. Είναι μήνυ ακρόαση επαναλαμβάνω και όπως γνωρίζετε κι εσείς είναι μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για την οποία εισηγητής είναι ο κύριος Νάγκη που είναι κοντά μας σήμερα και μετά τις τροπολογίες που υπέβαλαν οι συνάδελφοι στο σχέδιο έκθεση του κύριου Νάγκη, ο εισηγητής και οι σκιώδες αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται τις συμβαστικές τροπολογίες έτσι ώστε να εγκριθούν στην έκθεση στη συνεδρίαση με την έκθεση της ΛΥΜΠΕ στις 27 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή ακρόαση θα προσφέρει ε, μια πολύτιμη συνεισφορά έτσι ώστε να κλείσουμε αυτές τις συμβαστικές προτάσεις. Έχουμε μαζί μας αξιότιμους ε, εμπειρογνώμονες που γνωρίζουν καλά τον κλάδο των προτύπων σημειονότες. Να καλωσορίσω λοιπόν τον κύριο Τόγκενμπουργκ που είναι ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος στο γραφείο του Διευθυντή της Υπηρεσίας για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, τον κύριο Μάικλ Τόις που είναι επικεφαλής μονάδας για τα σχολεία ε, και την πολυγλωσία στην DG EAC, την κυρία Ζέτα Γεωργιάδου, που είναι αναπληρώτρια προϊσταμένη στη μονάδα για την πολιτική για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην DG, στην Γενική Διεύθυνση Just, και τη Γιάννα Μπαλαζόβα, που είναι ε, υπάλληλο ε, στην DG Dust, στο τμήμα για τη μη διάκριση και το συντονισμό για τα θέματα Ρώμα. Έχουμε επίση μαζί μα τον κύριο Λάιντεκερ, που είναι επικεφαλή γραμματεία από την Συμβουλευτική Επιτροπή για το Συμφωνία σύμβαση πλαίσιο για την ε, προστασία των εθνικών μειονοτήτων από το Συμβούλιο της Ευρώπης, την κυρία Χραμπανόβα, που είναι εκτελεστική διευθύντρια ε, της, του δικτύου έργο για τις οργανώσεις βάσης για τα δικαιώματα των Ρωμά και τον κύριο Μπουκοβόσκι, που είναι ο πληρεξούσιος της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβακίας για τις εθνικές μειονότητες, όπως επίσης και την κυρία Σλεζάκ, που είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τι καθημερινέ εφημερίδε ε, της σε μειονοτικές και περιφερειακές γλώσσες. Για να ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ζήσω καταρχήν ε, από τον κύριο Νάγκη, που είναι ο συγητής μας, να πει δύο λόγια και μετά θα ακούσουμε τους ομιλητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το γεγονός που συμμετέχετε κι εσείς ε, σε αυτό το θέμα που απασχολεί όλες τις εθνικές και περιφερειακές μειονότητες στην Ευρώπη. Ε, είναι ένα, μια έκτακτη εκδήλωση και αυτό εν ώψη του φακέλου που θα ψηφίσουμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε κάποια ελάχιστα πρότυπα για τις εθνικές μειονότητες και τις εθνοτικές ομάδες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω τη στήριξη και την πολιτική ε, βοήθεια όλων των εθνικών αντιπροσωπιών, των πολιτικών ομάδων και των συναδέλφων να σα υπενθυμίσω πως πάνω από 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες αυτή τη στιγμή ανήκουν ε, σε μειονότητες στη χώρα στην οποία κατοικούν. Και αν μπορούμε το έγγραφο αυτό να το υπερψηφίσουμε, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσει ένα κανονισμό ε, για τα ελάχιστα ε, δικαιώματα, όχι μόνο τα πολιτικά, θα τα αποκλείσουμε αυτά, αλλά για τα πολιτιστικά, τα εκπαιδευτικά, τα γλωσσικά κτλ. Νομίζω ότι θα έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, θα έχουμε στείλει το κατάλληλο μήνυμα και στα κράτη-μέλη, αλλά και σε ολόκληρη την εμφύλιο για το γεγονό πω η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ηγηθεί αυτή τη πολιτική. Ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ομιλητές σήμερα είναι εμπειρογνώμονες είναι εξαιρετικοί ομιλητές οι οποίοι θα μας δώσουν επιχειρήματα έτσι ώστε ε, να καταλάβουν όλοι πως αν εξασφαλίζουν τα δικαιώματα αυτών των ε, μειονοτήτων ε, θα αποκτήσουν και μεγαλύτερη ταύτιση με το εθνικό κράτος το οποίο ζουν. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Νάγκη και θα ήθελα χωρίς να καθυστερούμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Τόγκεμπεργκ καταρχήν όπως σας είπα από την υπηρεσία για τα θεομελιώδη δικαιώματα και έχετε μέχρι 7 λεπτά στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που καλέσατε την υπηρεσία μας σε αυτό το τόσο σημαντικό ε, θέμα θα ήθελα να απασχοληθούμε με τρία διαφορετικά θέματα. Πρώτον, αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, σχέση μεταξύ Συμβουλίου Ευρώπης και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τρίτον, σχέδιο έκθεσης, όπως αυτή τη στιγμή έχει το κείμενο μπροστά μας. Να ξεκινήσουμε καταρχήν με τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό το θέμα σήμερα γιατί εξαρτάται από το συνομιλητή κάθε φορά για να δούμε τι καθένα μας κατανοεί. Κάποιοι λένε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τίποτα να προσθέσει και τίποτα να πει για μειονότητες. Γιατί αυτό θα αποτελούσε καταπάτηση ε, της αρχής επικουρικότητας και της εκχώρησης αρμοδιοτήτων. Οπότε θα μας έλεγαν μην πείτε τίποτα. Άλλοι θα προσθέσουν πως ε, αυτή τη στιγμή είμαστε ε, το νέο έμβλημα των εθνικών μειονότητων γιατί υπάρχουν νέα ε, εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ξεπερνάν αυτά που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι και οι δύο απόψει είναι και σωστέ και λάθο. Καταρχήν για το πρώτο να σα πω θα εξαρτηθεί καταρχήν από το τι είδου διαχείρισης διαφορετικότητα έχει κάθε να μα κατά νου. Τι σημαίνει διαχείριση διαφορετικότητα. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να εξασκήσουμε σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Δηλαδή ποιο έχει δικαίωμα να μπει κανεί και να ζήσει στη χώρα σου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά να μπει και κυρίω. Ε, με τους μόνιμα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών ε, και βλέπετε ότι γίνεται και σε πολιτικό επίπεδο με τη συζήτηση για το προσφυγικό. Το δεύτερο είναι το κατά πόσο μπορούμε να ενσωματώσουμε ανθρώπους και πώς μπορούμε να επιτύχουμε την κοινωνική έντεξη με, καταπολεμώντας τις διακρίσεις και εδώ είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη που έχουν αρμοδιότητες και μάλιστα ε, πολλές. Και τρίτο είναι η διατήρηση. Δηλαδή ποιος έχει δικαίωμα συλλογικά να διατηρήσει μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να προσθέσει. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δίκιο όταν επαναλαμβάνει πως τα θέματα της περιφερειακής αυτονομίας, ε, της ε, ε, κοινωνικής διαστρωμάτωσης και όλων των συνοφών θεμάτων θα έπρεπε καλύτερα να τα αφήσει στα κράτη-μέλη. Τώρα, τι σχέση έχει και πώς σχετίζονται ε, το ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή αποτελεί το χρυσού κανόνα σε θέματα μειονοτήτων και θα παραμείνει νομίζω στο χώρο αυτό για τα επόμενα χρόνια. Και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που διαπιστώνω πως το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Νάγκη αναφέρεται στην κατευθυντήρια γραμμή 5 για τη νομική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης που εγκρίθηκε το 2005 όπου αναφέρεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσπαθήσει να μεταγράψει, να μεταφάρει, να μεταφέρει τις ε, υποχρεώσεις ε, διεθνούς δικαίου που έχει ε, καθορίσει το Συμβούλιο της Ευρώπης σε περίπτωση που εμπίπτουν στα πεδία νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δούμε λοιπόν την σύμβαση πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορεί κανείς να κατηγοριοποιήσει τις τρεις ομάδες εκεί τις διατάξεις. Καταρχήν έχουμε τις διατάξεις όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προσθέσει οτιδήποτε γιατί έχουν να κάνουν με περιφερειακή ε, αυτονομία, με συλλογική ταυτότητα, με πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε μειονετικές γλώσσες κτλ. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία να προσφέρει. Δεύτερον, Έχουμε τις άλλες διατάξεις, μια δεύτερη κατηγορία όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί δύναται να προσφέρει βοήθεια μέσω χρηματοδότησης, ε, ήπιων νομικών παρεμβάσεων κτλ. Δηλαδή, σα δώσω ένα παράδειγμα. Πώς μπορεί κανεί να σέβεται την ταυτότητα ατόμων που ανήκει σε εθνική μειονότητα. Ανήκουν σε εθνική μειονότητα. Και έχουμε και μια τρίτη κατηγορία διατάξεων στην ε, βασιπλαίσιο, όπου μπορεί ε, να ε, εγκρίνει νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, άρθρο 10, παράγραφος 3 της Συμφωνίας της Σύμβασης Πλαίσιο λέει πως αν κανείς συλληφθεί έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί για τα δικαιώματά του στην μητρική του γλώσσα. Στην ε, Οδηγία 64 που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αναφέρει στη μετάφραση και διερμηνία κατά τις ποινικέ διαδικασίες, μπορώ να σας πω πως το μόνο που κάνει είναι να μεταφέρει αυτές τις διεθνείς διατάξεις στο υπερεθνικό δίκαιο, έτσι ώστε να έχουν άμεση εφαρμογή και στο εθνικό δίκαιο. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα που δείχνει σε πόση μεγάλη ε, συνάφεια ε, είναι η νομοθεσία στο σημείο αυτό. Υπάρχουν λοιπόν κάποια θέματα όπου μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τις υποχρεώσεις που υπάρχουν στο διεθνές δίκαιο να τις μεταφέρει ε, στο δικό της, ε, στα δικά της νομικά εργαλεία έτσι ώστε να εφαρμοστούν και από τα κράτη-μέλη. Και να σας πω πως γενικότερα και βλέπετε πως προτιμώ να κατηγοροποιώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποιες διατάξεις που μπορούμε να διατηγοριοποιήσουμε και κάποιες παραγράφους ε, ε, τις οποίες θα χαρακτηρίσω ως ευχολόγιο. Μετά έχουμε και άλλες παραγράφους οι οποίοι έχουν συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τα κράτη-μέλη. Αυτά ε, αναφέρονται στην γνωμοδότηση που ετοιμάζει ο συνάδελφός σας και πρέπει να σου πω πως οι παράγραφοι αυτοί συνήθως συνδυάζονται, αλλά δημιουργούν και κάποιες δυσκολίες. Κοιτάξτε την παράγραφο 21 για παράδειγμα το Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει πω τα άτομα που ανήκουν στι εθνικέ μειονότητε έχουν το δικαίωμα να εκπαιδεύονται στη μειονοτική του γλώσσα. Νομίζω ότι ε, πολλά ζητάμε. Δεν μπορεί να επιβάλλει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να το προωθήσει, ναι. Να το διασφαλίσει, νομίζω, είναι τελείω εκτό πεδίου εφαρμογή ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επίσης, έχετε μια κατηγορία διατάξεων που απευθύνονται μόνο στα κράτη-μέλη ή μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέσσερις διατάξεις που απευθύνονται μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ θεωρώ πως δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κοιτάξτε την παράγραφο 22, όπου αναφέρεται πως η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει κάποιες μονάδες έτσι ώστε να εξασφαλιστούν τα, τα, τα μαθήματα σε μειονοτικές γλώσσες ε, στην διδακτέα ύλη στα σχολεία. Πολύ καλά όλα αυτά, αλλά πώς θα το εφαρμόσει. Συμπερασματικά λοιπόν θα πω το εξή. Λείπει κάτι από την έκθεση. Ε, βεβαίως μιλάμε για την θετική ένταξη στην έκθεση τη δική σας. Ναι, αλλά τι θα γίνει με την αρνητική ένταξη. Και τι είναι η αρνητική ένταξη. Είναι αυτή η οποία ε, απορρέει από τι τέσσερι βασικέ ελευθερίε. Δηλαδή, αν έχουμε ένα εθνικό σύστημα προστασία των μειονοτήτων σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και παρόλα αυτά οι κοινοτικέ διαδικασίε σα επιβάλλουν να ανοίξετε ε, τα πλεονεκτήματα που προσφέρετε στι μειονοτικέ ομάδε σε όλου του πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση, τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή. Μπορείτε να εξακολουθήσετε να προστατεύετε τι μειονότητε σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να το δώσετε. Και αυτό θα το τελευταίο τελευταίο που έχω να πω, πως δύο ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Καταρχήν, ο περιορισμό των ε, αρμοδιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερον το τεράστιο δυναμικό που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να, προσ... να επεκτείνουμε την προστασία που προσφέρουμε. αυτέ οι δύο διαστάσει πρέπει να τι δούμε και τι δύο πολύ σοβαρά. Διαφορετικά η δουλειά που θα κάνουμε δεν θα πάει αρκετά μακριά. Ευχαριστώ. Now to... Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα περάσουμε στον κύριο Λάιντεκερ. Μέχρι 7 λεπτά παρακαλώ. Ε, um, ε, my colleagues and myself are here to. Uh, συνάδελφοι και εγώ είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε μετά από τα όσα είπε ο κύριος Τόκενμπουργκ για να εξηγήσουμε ε, τις δράσεις της Επιτροπής που θα έπρεπε να είναι αποτελεσματικές όσον αφορά την προστασία των μειονοτήτων καθώς και τα όρια των αρμοδιοτήτων μας. Η βάση βεβαίως είναι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ανήκουν στις, σε μειονότητες. Είναι μια αρχή που αναφέρεται ρητά στο άρθρο 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόκειται για μια από τις ιδρυτικές αξίες της Ένωσης οι οποίες αντικατοπτρίζονται στον ε, χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι του χάρτη μεταφράζουν τις συγκεκριμένες αξίες σε άρθρα που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του χάρτη, απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση επί τη βάση της ένταξης σε μια εθνική μειονότητα, ενώ το άρθρο 2 του χάρτη ε, λέει ότι η Ένωση θα πρέπει να σέβεται τις πολιτιστικές, τις θρησκευτικές και τις γλωσσικές, τη γλωσσική μάλλον πολυμορφία. Ιδιαίτερα το δικαίωμα στην ε, μη διακρίση ε, θα πρέπει να μεριμνάται ε, από πλευρά τη Κομισιόν ώστε να γίνεται σεβαστό και να είναι εντεταγμένο στην νομοθεσία. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει γενικέ αρμοδιότητε να δράσει όσον αφορά τι μειονότητε. Το άρθρο 2 τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν μπορούν να σημεύσουν ω νομική βάση για νομοθετικά εργαλεία. Δεν υπάρχει δεν έχει η Κομισιόν αρμοδιότητες όσον αφορά τον ορισμό ε, του ε, καθεστώτος των μειονοτήτων, την αυτοδιάθεση αυτών ή το καθεστώς που καλύπτει τη χρήση περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών. Αυτά όλα εντάσσονται στις ευθύνες των κρατών μελών και ε, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συμμορφούνται με τη συνταγματικό του τα συνταγματικές υποχρεώσεις με το διεθνέ δίκαιο αλλά και να προβαίνουν σε απαραίτητα μέτρα ώστε να να προστατεύονται τα δικαιώματα των μειονοτήτων που ζουν στην επικράτειά τους και οι διεθνείς τους ε, ε, υποχρεώσει περιλαμβάνουν και αυτέ που απορρέουν από τα μέσα του Συμβουλίου τη Ευρώπη, όπω το πλαίσιο για την προστασία των, των μειονοτήτων ή το χάρτη για την προστασία των μειονοτικών γλωσσών. Ωστόσο, η συνθήκη δίνει κάποιε αρμοδιότητε στην Ένωση ώστε να αναπτύξει πολιτικέ που συμβάλλουν στην ε, προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τη Κομισιόν, η Κομισιόν ε, πρέπει να φτιάξει συντάξει τέτοιες πολιτικές που να εξασφαλίζουν το σεβασμό και την προώθηση των δικαιωμάτων που αφορούν ε, όλος ιδιαίτερος τους ανθρώπους που ανήκουν σε μειονότητες. Ε, δηλαδή, ε, μη διακρίσεις, καταπολέμηση της, του ρατσισμού και η προώθηση του πολιτιστικού, διαπολιτιστικού διαλόγου, της δημοκρατικής συμμετοχής και η στήριξη των δράσεων των κρατών μελών, όπω η προώθηση της πολυγλωσσίας και η χρήση, της χρήσης μάλλον των μειονοτικών γλωσσών σημαντικό στοιχείο κατά των διακρίσεων είναι η περίφημη απόφαση να ε, καταπολεμηθεί ο ρατσισμός και οι διακρίσεις με βάση το ποινικό δίκαιο. Ε, οπότε ε, καταδικάζεται ο λόγος μίσους, ε, hate speech, είτε αφορά χρώμα, είτε εθνικότητα, είτε θρησκεία, είτε οτιδήποτε άλλο. Η οδηγία της Κομισιόν επίσης καταδικάζει τον λόγο μίσους, απαγορεύοντας την χρήση του για οποιοδήποτε θέμα, εθνικότητα, φιλή, χρώμα, και τα, θρησκεία κτλ. η Κομισιόν λοιπόν πρέπει να φροντίσει ώστε τα κράτη-μέλη να συμμορφούνται προς αυτήν την ε, οδηγία. Με βάση την αναθεώρηση της οδηγίας τώρα περί των μέσων μαζικής ενημέρωσης καλύπτεται και εκεί το θέμα της καταπολέμησης των διακρίσεων για οποιοδήποτε λόγο. Επιπλέον η Κομισιόν έχει λάβει μια σειρά μέτρων ώστε να βοηθήσει να εξασφαλιστεί πως το μίσος και η μη ανοχή καταπολεμώνται επί τόπου. Όπως γνωρίζει η Κομισιόν το 2016 συμφώνησε σε ε, ε, για έναν ε, κώδικα διοντολογίας ε, που στόχο έχει να αντιπαρατεθεί στο λόγο μίσους επιγραμμικά. Δηλαδή αυτό έχει γίνει δεκτό από το Instagram και διάφορες άλλες πλατφόρμες του, του διαδικτύου. Η πρόσφατη αξιολόγηση δείχνει πως αυτή η οδηγία έχει αφαιρέσει 70% του λόγου μίσους από το τα τελευταία χρόνια ε, η Κομισιόν έχει ε, υποστηρίξει ΜΚΟ ε, που παρακολουθούν το τι συμβαίνει, παρακολουθούν το λόγο μίσους online ώστε να ε, παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Επίσης έχουμε φτιάξει μια ομάδα υψηλού επίπεδου που συμμετέχουν όλα τα κρατημέλη, διεθνεί οργανισμοί και βασικές οργανώσεις ε, των πολιτών ώστε να εντοπίζουν συγκεκριμένους, ε, συγκεκριμένα είδη μη ανοχής και στόχος είναι να δούμε πώς θα βελτιώσουμε και την κατάσταση, πώ θα διώξουμε το, τις περιστάσεις ε, μάλλον τα περιστατικά μίσους ε, και πώς θα βοηθήσουμε τα θύματα. Επίσης παρέχουμε στηρίξη μέσω του προγράμματος δικαιωμάτων του πολίτη και βοηθάμε την κοινωνία των πολιτών αλλά και τα κρατημέλη ώστε να καταπολεμήσουν ε, τον ρατσισμό και το λόγο ε, μίσους. Ε, συγκεκριμένες μορφές μη ανοχής, μη ανεκτικότητας επίσης κατά των τσιγκάνων. Ε, ένας άλλος τομέας όπου η Κομισιόν ε, δρά για τα δικαιώματα ανθρώπων που ανήκουν στις μειονότητες είναι η πρόθεση της δημοκρατικής συμμετοχής. Είπα ε, σύμφωνα μάλλον με την έκθεση του 2017, είναι προτεραιότητα της Κομισιόν να προωθήσει την ε, συμμετοχή των κινούμενων πολιτών στις χώρες υποδοχής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ομάδες που δεν εκπροσωπούνται παρκώς. Είναι στόχος ε, η ευρεία συμμετοχή στις ευρωεκλογέ. Είναι κοινή όμως αυτή η ευθύνη και με τα κράτη-μέλη και βοηθάμε τα κράτη-μέλη ώστε να διευκολύνουν τη συμμετοχή στις εκλογές όλων των Ευρωπαίων πολιτών και μάλιστα να αυξηθεί η συμμετοχή των ε, ομάδων που δεν ε, εκπροσωπούνται αρκετά. διερευνούμε πώς ε, με τις καλύτερες πρακτικές θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τη συμμετοχή των λιγότερων εκπροσωπούμενων ομάδων και τον Νοέμβριο φέτος θα αφιερώσουμε συνέδριο στο θέμα της δημοκρατίας όπου θα, ε, θα συζητηθεί και η δημοκρατική συμμετοχή των ε, λιγότερων εκπροσωπούμενων ομάδων όπως οι ομάδες μειονοτήτων. Συμμετέχουμε και σε διάφορα project που, προσέχουν, που προωθούν τη συμμετοχή των κινούμενων πολιτών στις δημοκρατικές δημοκρατικές διαδικασίες. Θέλουμε να προωθήσουμε την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία με αυτούς τους γενικούς στόχους. Αν μου επιτρέπετε τώρα να δώσω το λόγο στη συνάδελφο που θα εστιάσει περισσότερο στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Σας ευχαριστώ. Όπως μόλις ακούσατε, όσον αφορά την εντολή και τις αρμοδιότητες, ε, έχουμε διάφορα μέσα ε, στη διάθεσή μας για να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις. Εγώ θέλω να μιλήσω για την οδηγία για τις ε, φιλετικές για την, στη φιλετική ισότητα. Το 2015 η Κομισιόν ξεκίνησε την πρώτη διαδικασία κατά παράβαση για θέμα διακρίσεων επί εθνική, βάσης. Ήταν οι διακρίσεις που υφίστανται τα παιδιά Ρωμά στην, ε, μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους στην Τσεχία ε, και ξεκίνησε και μια διαδικασία κατά παράβαση κατά της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας για τους ίδιους λόγους ε, στη συνέχεια. Ω θεματοφύλακα των συνθήκων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πολύ σοβαρά λαμβάνει υπόψη αυτά τα θέματα, ειδικά όταν πρόκειται για παραβάση, παραβίαση μάλλον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε, ε, τώρα, όσον αφορά τις διαδικασίες κατά παράβαση, θα θέλω να τονίσω ότι στόχος δεν ήταν να τιμωρήσουμε τα κρατημέλη, αλλά σε στενή συνεργασία να διορθώσουμε την κατάσταση αυτή, δηλαδή να εξασφαλίσουμε πως τα παιδιά Ρώμα θα έχουν την ίδια πρόσβαση σε ποιοτική ε, και καθολική παιδεία όπως οποιαδήποτε άλλα παιδιά στις χώρες αυτές. Τώρα, όσον αφορά τους Ρωμά, η κατάσταση είναι περίπλοκη, ιδιαίτερα περίπλοκη. Αναφέρομαι ειδικά στη Ρωμά, στους Ρωμά, γιατί είναι η μεγαλύτερη μειονότητα της Ευρώπης. Ε, εκτιμάται ότι είναι περίπου 10 με 12 εκατομμύρια και στις χώρες διεύρυνσης. Ε. Όπως είπα, είναι περίπλοκη η κατάσταση και οι λύσεις δεν είναι απλές, καθώς δεν πρόκειται μόνο για διακρίσεις, αλλά και για κοινωνική και οικονομική περιθωριοποίηση. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν σε πολύ ε, άσχημες ε, συνθήκες. Τον 21ο αιώνα έχουμε μέσα στην επικράτειά μας ε, χώρες όπου οι Ρωμά δεν έχουν πρόσβαση καν σε πόσιμο νερό ή σε βασικές ε, υπηρεσίες. Ε, τώρα μπορεί να μην το μπορείτε καν να το φανταστείτε, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτό επηρεάζει την υγεία τους, τα παιδιά συχνά πηγαίνουν σε σχολεία για παιδιά με ειδικέ ανάγκες ενώ είναι απόλυτα υγιή και αυτό γιατί δεν μιλούν τη γλώσσα της χώρας ε, όπου βρίσκονται ε, όταν ε, φτάνουν την ηλικία των 6 και δεν έχουν τις δεξιότητες που αναμένεται να έχουν τα παιδιά της ηλικία τους. Είναι πολύ περίπλοκη η κατάσταση λοιπόν, οι λύσεις δεν είναι εύκολες και η κατάσταση αυτή, καθώς και οι διακρίσεις κατά τον Ρωμά, είναι πολύ διαδεδομένες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό για... υπάρχουν δύο λόγοι και δύο βασικοί στόχοι που η Ευρώπη ε, ασχολήθηκε με αυτό το θέμα σαν προτεραιότητα από το 2010. Έκτοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτιάξει πολιτικά μέσα, ε, στο οποίο αναφέρθηκε και η συνάδελφος Ζέτα, παρακολουθεί την πρόοδο που έχουν ε, σημειώσει τα κράτη-μέλη έκτοτε. Δεν είναι τόσο γρήγορες οι εξελίξεις όσο θα θέλαμε, αλλά κάποιες βελτιώσεις είναι ήδη ορατές. Αυτή τη στιγμή ε, διεξάγουμε ε, εις βάθος ε, αξιολόγηση του βασικού μέσου πολιτικής που φτιάχτηκε το 10 για την, την εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών για τους Ρωμά. Διάφορα κράτη-μέλη συνέβαλαν στην αξιολόγηση μέσω της online διαβούλευσης και τα πορίσματα που θα δημοσιευθούν πριν το τέλος του έτους, τον Νοέμβριο δηλαδή υπολογίζουμε παρακολουθούμε την πρόοδο των κρατών μελών, γιατί εδώ θέλω να καταστήσω σαφέ ότι η βασική ευθύνη για την ένταξη των περιθωριοποιημένων πληθυσμών βαραίνει τα κρατημέλη. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια αρμοδιότητα, αλλά περιορισμένη, γιατί μιλάμε για Ευρωπαίου πολίτες, αλλά βασική κύρια ευθύνη ε, βαραίνει, όπω είπα, τα ε, κρατημέλη. μελη η πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη-μέλη παρακολουθείται σύμφωνα, μάλλον υπό το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 και έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες κατά παράβαση. Μίλησα για φιλετική ισότητα, αλλά άλλη σημαντική οδηγία είναι η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση που υιοθετήθηκε το 2000 και μιλά για διακρίσεις επί άλλης βάσης, αλλά περιορίζεται στην απασχόληση. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την οδηγία της για μια, στηρίζει μάλλον την πρότασή της για μια νέα οδηγία που θα επεκτείνει τις αρμοδιότητες και δεν θα περιορίζεται μόνο στην απασχόληση. Θα σταματήσω εδώ και βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Okay, Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάποιον ακόμα εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα πω δύο λόγια για το θέμα της παιδείας και του πολιτισμού. Είστε ο Μάικλ Τόις, μάλιστα. Νομίζω ότι λείπετε, αλλά βλέπω πώς είστε εδώ. Σας παρακαλώ πάντως να είστε σύντομος, γιατί έχουμε και πολλούς ακόμα ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ σχετικά με τα θέματα παιδείας και πολιτισμού, τα οποία αναφέρονται και αυτά στην έκθεση, να σας πω πως η νομική βάση στην οποία βασιζόμαστε είναι το άρθρο 165 και το άρθρο 167 της συνθήκης, τα οποία απερίδραστα δηλώνουν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και όπου χρειάζεται να προσθέτει και να ενισχύει τη δράση τους. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να προωθήσουμε και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν πολιτικές, γνωρίζοντας βέβαια πως η ευθύνη παραμένει στα χέρια των κρατομελών για τα θέματα αυτά. Οπότε με αυτή τη βάση έχουμε ένα είδος πολιτικής συνεργασίας και προς αυτή την κατεύθυνση χρησιμοποιούμε και τις δικές μας ε, δυνατότητες. Ε, μίλησε για το χρυσού κανόνα ο κύριο Τόκενμπουργκ και νομίζω ότι όντω έχουμε συνεργαστεί πολύ με το Συμβούλιο της Ευρώπης στο σημείο αυτό. Έχουμε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Ευρωπαϊκές Μειονοτικέ Γλώσσες. Είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που έχουμε ε, για την παιδεία στην, στο διεθνή χώρο και έχουμε επίσης αυτή τη χάρτα που έχει η υιοθετηθεί από τα περισσότερα κράτη-μέλη. Έχουμε και στο κράτη το Κέντρο για τι Ευρωπαϊκές Γλώσσες και μέσω του Συμβουλίου τη Ευρώπη προσπαθούμε να προωθήσουμε και κάποια θέματα. Στην πράξη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμεί προωθούμε την ε, εκμάθηση γλωσσών και πρόσφατα καταθέσαμε και μία πρόταση για την εκμάθηση γλωσσών που λαμβάνει υπόψη την ε, ε, πληθώρα γλώσσεων που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προωθούμε λοιπόν όχι μόνο τι επίσημε γλώσσε κάθε κράτου μέλου, αλλά και συζητάμε το θέμα αυτό με τα κράτη-μέλη, προωθούμε και τη διδασκαλία και εκμάθηση όλων των γλωσσών που υπάρχουν μέσω συνεργασίας αλλά και μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Το πιο σημαντικό είναι το Erasmus Plus και στα πλαίσια του Erasmus προωθούμε όλες τις γλώσσες, την εκμάθηση όλων των γλωσσών. Έχουμε πολλά project για την εκμάθηση που συμπεριλαμβάνουν και γλώσσες μειονοτικές. Βεβαίως αυτό δεν ε, σημαίνει πως θα προκρίνουμε μόνο τις επίσημες γλώσσες, αλλά να σας πω πως τον Ιούνιο πήγα ε, στην ε, δική σας ομάδα ε, για τις ε, μειονοτικές γλώσσες και παρουσίασα τις προσπαθίες μας εκεί, να σας πω πως είναι ένα θέμα στο οποίο κάνουμε ό,τι μπορούμε και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Υπάρχουν οι ευκαιρίες αυτές και βεβαίως η νομική αρμοδιότητα αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια των κρατών μελών. Αλλά ανταλλάσσουμε τις βέλτιε πρακτικέ, έτσι ώστε η, η πολυμορφία γλωσσών που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να προωθηθεί στο μέτρο του δυνατό. Σα ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι της έκθεσης για την ε, πολυγλωσσία, οπότε σας ευχαριστώ που μας δώσετε αυτές τις επιπλέον πληροφορίες. Θα μπορέσουμε τώρα να προχωρήσουμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Μάρκο Λάιντεκερ. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Είναι και χαρά αλλά και τιμή. Μεγάλη τιμή. Που σας παρουσιάζω ένα θέμα το οποίο αποκτά όλο και περισσότερη απήχηση στην Ευρώπη. Προστασία των εθνικών μειονοτήτων λοιπόν. Να ασχοληθώ με τα θέματα. Πρώτον, ο ρόλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πολύ χαρά άκουσα να αναφέρεται επανειλημμένα το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν θα τα πω όλα βέβαια, αλλά να πάω λίγο περισσότερο σε βάθος. Και επίσης ε, θα ήθελα να μιλήσω για τη Συμφωνία Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων. Πώς λειτουργεί, ποια είναι η δομή της και ίσως πιο σημαντικό για τις συζητήσεις σας, η συνεργασία με μια σειρά άλλα μέσα για την προστασία των μειονοτήτων. Τώρα το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν θα σας εκπλήξει ότι έχουμε ασχοληθεί εδώ και πολλά χρόνια με το θέμα αυτό. Οι ιστορικοί λένε ότι η πρώτη φορά που αναφέρθηκε η ανάγκη προστασίας ε, των εθνικών μειονοτήτων το 1949 ήταν κατά την πρώτη χρονιά λειτουργίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για πάρα πολλά χρόνια το είχαμε αυτό το θέμα στην ημερήσια μας διάταξη και το 1993 μετά την κατέρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την ε, έκρηξη των ε, συγκρούσεων στην πρώην Ιουγκοσλαβία σε εθνοτική βάση το θέμα επανήλθε πολύ στην επικαιρότητα και το 1993 υπήρξε μια συνάντηση κορυφή όπου δημιουργήθηκαν δύο μέσα. Το πρώτο είναι λοιπόν αυτή η συμφωνία η σύμβαση πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μητών και, το, και η Ευρωπαϊκή Χάρτα για τις περιφερειακές και μελλοντικές γλώσσες. στι 19 και 20 Ιουνίου τρέχοντος είχαμε λοιπόν 20 ε, χρόνια από την έναρξη ισχύω αυτών των δύο συμβάσεων. Κάναμε μια αρκετά μεγάλη διάσκεψη για δύο μέρες με πολλούς υπουργού στο Στρασβούργο, κάτι που δείχνει ότι και τα δύο αυτά μέσα εξακολουθούν να είναι ενεργά. Έχουμε λοιπόν την επιτήρηση, έχουμε τη δημιουργία προδιαγραφών μέσω αυτών των δύο συμβάσεων, αλλά επιπλέον, συχνά και όλο και περισσότερο, το Συμβούλιο της Ευρώπης λοιπόν καλείται να αναλάβει στοχευμένες δράσεις συνεργασίας για να στηρίξει τα κράτη-μέλη της. Συγκεκριμένα φέτος, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει δώσει συμβουλές για θέματα νομοθεσίας για τις εθνικές μειονότητες στην Αλβανία, την Αρμενία και την Ουκρανία. Συχνά λοιπόν, βεβαίως, για τα θέματα αυτά συνεργαζόμεθα με το γραφείο του ΙΠΑ του αρμοστή για τις εθνικές μειονότητες στη Χάγη. Και βεβαίως, εφόσον εκπροσωπώ το Συμβούλιο της Ευρώπης, πρέπει να αναφερθώ και στην ε, Επιτροπή της Βενετίας. Από το 1999 έχει εγκρίνει μια σειρά από γνωμοδοτήσεις για συνταγματικά και θεσμικά σχέδια νόμου για τα δικαιώματα των μειονοτήτων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Να αναφέρω ορισμένες. Βοσνία Σεβοβίνη, Κροατία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ρουμανία και Ουκρανία. Που καλύπτουν πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων η χρήση των ε, γλωσσών στην δημόσια επικοινωνία, μειωνοτικέ γλώσσες στην ε, παιδεία, ακόμη και το καθεστώς των μειωνοτικών γλωσσών και το καθεστώς των ε, τοπικών πληθυσμών. Να προσπαθήσω να συμβάλλω στη συζήτησή σας για το σχέδιο ψηφίσματος. ενημερώνοντάς σας για τις δραστηριότητες της ε, Σύμβασης Πλαίσιο. Να θυμίσω ότι η Σύμβαση αυτή είναι το μόνο νομικά δεσμευτικό πολυμερές μέσο που ασχολείται αποκλειστικά με την προστασία των εθνικών μειονοτήτων. Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη σύναψή της το 1999 είναι ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα γιατί η επικύρωσή της καλεί τα κράτη να σεβαστούν έναν εκτεταμένο κατάλογο μειονοτικών δικαιωμάτων. Μεταξύ άλλων αναφέρουν το δικαίωμα ελεύθερης χρήσης και, και χωρίς καμία παρέμβαση τη μειονοτική γλώσσα στην ιδιωτική ζωή, τη δημόσια ζωή, γραπτός και προφορικός. Το δικαίωμα να έχει κανείς ε, μικρά ονόματα και επώνυμα σε αυτή τη γλώσσα το δικαίωμα να δημιουργεί και να διαχειρίζεται ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και το δικαίωμα εκμάθησης αυτών των μειωνοτικών γλωσσών. Επιπλέον η Σύμβαση επιβάλλει στα κράτη την υποχρέωση να προωθήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να μπορούν να ασκηθούν αυτά τα μειωνοτικά δικαιώματα, το οποίο σημαίνει δυνατότητες για εκπαίδευση ε, διδασκόντων, πρόσβαση σε σχολικά εγχειρίδια, και άλλα. Βεβαίως η σύμβαση πλαίσιο δεν είναι συνθήκη που τυφλά προωθεί αυτά τα δικαιώματα. Λαμβάνει υπόψη και άλλα σημαντικά συμφέροντα συνολικά της κοινωνίας. Θέλει απλώς να βοηθήσει τα κράτη να διατηρηθεί μια ενοποιημένη κοινωνία όπου να γίνονται αποδεκτά τα άτομα που προέρχονται από εθνικές μενότητε και μπορούν να ευημερούν πέρα από την εισαγωγή αυτών των δικαιωμάτων στην, ε, στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών και πέρα από τις συμβουλές που δίνει για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών, επιτηρεί επιπλέον ενεργά την εφαρμογή των υποχρεώσεων αυτών, δίνει πενταετής γνωμοδοτήσεις από μια ανεξάρτητη και αμερόληπτη συμβουλευτική επιτροπή και κατόπιν υπάρχουν ψήφισμα υπάρχουν και ψηφίσματα που εγκρίνονται από τι Επιτροπέ Υπουργών του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Μέχρι στιγμή, 39 κράτη-μέλη έχουν υπογράψει και επικυρώσει αυτή την σύμβαση και με μία, μετά από μια ειδική συμφωνία με την αποστολή των ΗΠΑ στο Κοσφοπέδιο, εφαρμόζεται και στο Κοσφοπέδιο. Τα 24 κράτη-μέλη από τα 39 αυτά είναι και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, μεν δεν είναι ενωσιακό μέσο, αλλά επειδή 24 από τα 28 κράτη-μέλη είναι συμβαλόμενα και σε αυτή τη σύμβαση παρέχει την πιο εκτεταμένη προστασία των ε, ε, εθνικών μειονοτήτων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον 16 κράτη-μέλη της Ένωσης επικύρωσαν και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις ε, περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες. Τώρα αν θα είχα λίγα λεπτά παραπάνω θα αναφερθώ σε μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της σύμβασης πλαίσιο και γενικά της προστασίας των εθνικών μειοτήτων που μπορεί να σας βοηθήσουν στις περαιτέρω συζητήσεις σας για το σχέδιο ψηφίσματος. Πρώτον και ιδιαίτερο σημαντικό. Δεν υπάρχει διεθνώς γενικά αποδεκτός ορισμός του τι αποτελεί εθνική μειονότητα. Οι απόψεις για το τι αποτελεί εθνική μειονότητα αποκλίνουν πολύ. Αυτό εξηγεί γιατί είναι τόσο διαφορετικοί οι εθνικοί ορισμοί που ακολουθούν ε, τα συμβαλόμενα κράτη. Η σύμβαση πλαίσιο δεν περιέχει ένα τέτοιο ορισμό. Αλλά δεν είναι μόνη της. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο κείμενο για το τι σημαίνουν οι εθνικές μειονότητες ούτε από τα Ηνωμένα Έθνη ούτε από τον ΟΑΣΕ. Οπότε, με βάση την σύμβαση πλαίσιο, τα κράτη-μέλη καθορίζουν το πεδίο εφαρμογή αυτού του μέσου. Ωστόσο, η Συμβουλευτική Επιτροπή που είναι τμήμα της σύμβασης μπορεί να θέσει πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις, ούτω ώστε να μην ε, εξαιρούνται διάφορες ομάδες από το πεδίο εφαρμογή αυτής της ε, σύμβασης με αυθαίρετο τρόπο και πολλές φορές ε, τα σχόλια αυτής της ε, Συμβουλευτικής Επιτροπής οδηγούν σε ένα διάλογο όχι μόνο μεταξύ αυτών των δύο μελών, δηλαδή του κράτους μέλους και της Συμβουλευτικής Επιτροπής, αλλά και εντός του κράτους μέλους. Και χάρη σε τέτοιο διάλογο, η έλλειψη ορισμού δημιουργεί την αναγκαία ευελιξία του μέσου αυτού. Κάτι που βεβαίως βοηθάει την προστασία των εθνικών μειονοτήτων. Η έλλειψη ορισμού μπορεί να οδηγήσει σε ένα άλλο ε, σημαντικό στοιχείο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων είναι δηλαδή το δικαίωμα αυτοκαθορισμού. Το αναφέρει συγκεκριμένο άρθρο. Ο αυτοκαθορισμός είναι σημαντικό ανθρώπινο δικαίωμα και η ευρωπαϊκή ιστορία καταδεικνύει το τι κίνδυνοι προκύπτουν όταν ε, κάποιος άλλος, για παράδειγμα ένα κράτος, επιβάλλει τον καθορισμό μιας ε, εθνικής μειονότητας. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να ασκείται καλό προαίρετα, αναφέρει η Σύμβαση. Και να αναφέρω κάτι ακόμη. Το κείμενο λέει δηλαδή, συγκεκριμένα 3-1 δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε, ούτε υπονοεί ότι ένα οποιοδήποτε άτομο έχει αυθερέτως και υποκειμενικά το δικαίωμα να επιλέξει σε ποια εθνική μειονότητα ανήκει. Αυτό έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά του ατόμου. Και αυτό με φέρνει σε ένα τέτοιο χαρακτηριστικό αυτής της σύμβασης. Η σύμβαση αυτή δεν είναι μέσο καταπολέμησης των διακρίσεων μόνο, αποκλειστικά. Είπαμε πολλά για την εντολή κατά καταπολέμηση των διακρίσεων που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το μέσο όμως είναι πολύ ευρύτερο. Και παραθέτω και πάλι για να καταλάβετε σαφώς τι εννοώ. Στο άρθρο 4.2 λέει ότι τα συμβαλόμενα μέρη, εάν χρειάζεται, δεσμεύονται να υιοθετήσουν τα αναγκαία μέτρα ούτω ώστε σε όλου του τομεί τη πολιτική, οικονομική και πολιτιστικής ζωή να υπάρχει πλήρης ισότητα μεταξύ των ατόμων που ανήκουν σε μια εθνική μειονότητα και των ατόμων που ανήκουν στην πλειονότητα. Και κατόπιν, πολύ βασικό, τα μέτρα αυτά δεν θα θεωρηθούν διακρίσεις. Δεν είναι λοιπόν μόνο μέσο καταπολέμησης των διακρίσεων, είναι πολύ ευρύτερο. Ίσως αυτό θα θέλατε και εσείς να το λάβετε υπόψη όταν θα συζητήσετε το ψήφισμα. Η σύμβαση πλαίσιο όμως ε, δεν λειτουργεί εν κενό. Έχουμε το 92 τη διακήρυξη των ΟΕΕ Εθνών για τα άτομα που συμμετέχουν, που ε, είναι μέλη εθνικής, θρησκευτική ή πολιτιστικής μειονότητας που παριλαμβάνουν παρόμοιες διατάξει. Και τα δύο αυτά μέσα, η διακήρυξη των ΟΕΕ και η σύμβαση πλαίσιο, είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας ε, σταδιακής εγκατάλειψη τη νομική προσέγγιση που υπήρχε και κυριαρχούσε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που θεωρούσε ότι η προστασία των μειονοτήτων μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με γενικά νομικά μέσα για την ισότητα όλων των πολιτών. Έχουμε λοιπόν ε, ξεπεράσει αυτό το πλαίσιο. Όμως ε, την τελευταία δεκαετία διαπιστώσαμε ότι τα θετικά μέτρα από το κράτος θα είναι αναγκαία για να υπάρξουν για να υπάρξει αναγκαία προστασία των ε, μειονοτήτων. Με συγχωρείτε που μακρηγορώ και συγγνώμη. Αλλά το έκανα αυτό για να συμβάλλω όσο μπορώ πιο ουσιοδός στην εργασία σας. Όπως ξέρετε σε πολλά κράτη-μέλη τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων ε, υφίστανται διάβρωση και μειώνονται. Άρα η προσπάθειά σας μπορεί να είναι δυσχερής και ελπίζω η συμβολή μου να διευκολύνει λίγο την ε, προσπάθειά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι εξαιρετική η παρουσίαση που κάνατε για τη σύμβαση πλαίσιο. Βεβαίω, για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράγματα είναι τελείω διαφορετικά. Εμεί δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την άγουσα τη ε, σύμβαση. Είναι ακόμα πιο περίπλοκη η δική μα κατάσταση με τι μειονότητε και γι' αυτό είναι τόσο διαφορετικά τα όσα επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει λοιπόν μια σφαιρική προσέγγιση που να μπορούμε να, συνολική που να μπορούμε να ε, ακολουθήσουμε και αυτό έχουμε όλες τις διαφορετικές εκθέσεις οι οποίες εστιάζουν σε διαφορετικούς τομείς κάθε φορά. Είναι όμως πολύ καλό να ακούει κανείς τι κάνει το Συμβούλιο της Ευρώπης γιατί νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι από τη βασική σας κληρονομιά και είναι και πολύ ουσιαστικό για την προσπάθεια που κάνουμε στη δική μας έκθεση. Θα περάσουμε λοιπόν κατευθείαν στην εκτελεστική ε, διευθύντρια της ΕΡΓΟ που είναι η Ευρωπαϊ... το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Οργανώσεων Βάσης για τους Ρωμά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και για την πρόσκληση που απευθύνονται να είμαι εδώ σήμερα. Εκ μέρους της ΕΡΓΟ λοιπόν ήθελα να χαιρετήσω αυτή την προσπάθεια που κάνει για ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ελάχιστα δικαιώματα και τις μειονότητες στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζονται ως μειονότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι Ρωμά και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός αυτής. Είμαστε ένα δίκτυο των ε, οργανώσεων βάσης των Ρωμά για να σας παρουσιάσουμε ε, την καθημερινότητά μας και τι κάνουν οι ΜΚΑ ομικρών στις καθημερινές τους προσπάθειες. Έχουμε 35 ενώσεις που βρίσκονται και στην Ευρώπη και στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Ουκρανία και στην Τουρκία και χαιρόμαστε που η ευρωπαϊκή κληρονομιά είναι τόσο πλούσια σε επίπεδο μειονοτήτων και χαιρόμαστε που προσφέρουν και οι Ρωμά. Η, η προστασία των μειονοτήτων όμως και τα κριτήρια της Κοπεχάγης δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο από όλους και δεν προστατεύονται πάντοτε. Υπάρχει μια διαφορετική εφαρμογή γιατί καταρχήν ποιο αποτελεί τη μειονοτική ομάδα και πολλές φορές οι κυβερνήσεις κάνουν και μια διάκριση και έχουμε εθνικές, εθνοτικές, θρησκευτικέ και λοιπές μειονότητες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε καταρχήν πώς θα τις ορίσουμε τα δικαιώματά τους και να εξασφαλίσουμε και την προστασία τους και κυρίως κατά των διακρίσεων και όλων των μορφών ρατσισμού. Να σας δώσω μια γρήγορη επισκόπηση για το που αναγνωρίζεται ο Ρωμός μειονότητα και για τους Ρωμά να σας πω πως τα πρότυπα είναι απολύτως απαραίτητα, αναγνωρίζοντας εθνική μειονότητα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη που έχουν και τι μεγάλες συγκεντρώσει πληθυσμού. Εκεί ε, ε, έχουν βασικά δικαιώματα, για παράδειγμα στην ε, Τσεχία, που έχουν και πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Όμως η επίσημη πολιτική δεν έχει πετύχει να βελτιωθούν σημαντικά τα προβλήματα περιθωριοποίησης, επιθέσεων, εκφοβισμού που αντιμετωπίζουν στις χώρες αυτές οι Ρωμά. Ιταλία, Γαλλία, ε, Ισπανία και Ελλάδα, πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δεν θεωρούνται εθνική μειονότητα εκεί η Ρώμα από το κράτο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ορίζεται νομικά αυτό ο όρο εθνική μειονότητα. Όμω οι αρχέ χρησιμοποιούν τον βασικό. Ε, το βασικό ορισμό που είναι η Ρωμά, η Τσιγκάνη και η ε, οδηπόροι ε, και αυτούς τους ορισμούς χρησιμοποιούν ε, ευρύτερα. Έχουν έναν ορισμό που περνά από τη βολή των, ε, της Ιταλίας, αλλά δεν έχει υπερψηφιστεί ακόμα. Αναγνωρίζονται στην Γερμανία, αλλά μόνο αυτοί οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι και όχι αυτοί που είναι ταξιδιώτες. Αναγνωρίζονται λοιπόν στην Γαλλία. Η κατάσταση είναι διαφορετική στην Αυστρία που από το 1993 αναγνωρίζεται ως εθνική μειονότητα αλλά όταν λέμε εθνική ομάδα περιορίζουμε εδώ στους αυτόχθονες Ρωμά και στους Σύντι οι οποίοι ζουν από το 15ο αιώνα στη χώρα αυτή. Οι κοινότητες Ρωμά που έχουν μεταφερθεί από τη δεκαετία του 60 μετακινηθεί προς την Αυστρία δεν αναγνωρίζονται παρόλο που αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα των Ρωμά που διαβιούν στην Αυστρία σήμερα. Η Ιρλανδία αναγνωρίζει και τους αναγνωρίζει ως ταξιδιώτες, ως travelers από πέρυσι. Οι Ρωμά όμως δεν αναγνωρίζονται ως Ρώμα. Να σας πω λοιπόν πως στη Φιλανδία αναγνωρίζονται από τότε ε, που ε, ισχύει το συγκεκριμένο σύνταγμα και θεωρείται εθνική μειονότητα. Αυτά σας τα παρουσιάζουν στοιχεία από ε, τον Κέντρο Παρακολούθησης των Ρωμά που χρησιμοποιούμε για να ε, δούμε πώς εξελίσσονται οι πληθυσμοί Ρωμά στην Ευρώπη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι είναι ε, κοινά. Δηλαδή δεν υπάρχουν ε, κονδύλια για να ενταχθούν οι Ρωμά σε πολλά κράτη-μέλη και πολλές φορές και οι θεσμοί που εκπροσωπούν τους Ρωμά δεν μπορούν να τεκμηριώσουν τις διακρίσεις που υφίστανται. Κάποια κράτη-μέλη έχουν δημιουργήσει τους θεσμούς που τους επιτρέπει σε εθνικό επίπεδο να καταπολεμούσουν τα κηρύγματα μίσους και να σας πω το εξή. Οι Ισπανικές περιφέρειες αυτή τη στιγμή έχουν ειδικό εισαγγελέα ε, που είναι ε, ε, ειδικό και εξειδικευμένος σε θέματα κηρύγματος μίσους και διακρίσεων κατά των διακρίσεων για τους Ρωμά. Αλλά δεν αναγνωρίζονται αυτά νομοθετικά και πολλές φορές οι θεσμοί δεν αναγνωρίζουν το ότι οι Ρωμά αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα. Πιστεύω λοιπόν πως γενικά οι πολιτικές δομές σε όλες τις χώρες ε, είναι αρκετά έθραυτες, γιατί πολλές φορές εξαρτώνται και από το κοινωνικό κλίμα το οποίο υπερισχύει σε κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Να σας πω λοιπόν πως το πρόβλημα είναι πως για τις μειονότητες Ρωμά δεν υπάρχει κάποιο κράτος ε, ε πατρίδα το οποίο να του στηρίζει. Ε, πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε και τα ελάχιστα πρότυπα για την αναγνώριση και την προστασία αλλά και την προστασία της γλώσσας τους. Αποτελεί η δικλίδα ασφαλείας Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει ελπίδες και όπως λέει και το ψήφισμα ε, ε, από το 2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από την έκθεση του 2017 πρέπει να σας πω πως διαπιστώνουμε πως η κατάσταση των Ρωμά χειροτερεύει. Χρειάζεται επίγουσα δράση για να αντιστρέψει την κατάσταση αυτή της αιώνιας, ε, μάλλον της εδώ και αιώνες περιθωριοποίησης των Ρωμά, της Διάκριση αυτή κατά των εθνικών αυτών μειονοτήτων. Να σας πω λοιπόν πως έχουμε πάρα πολλές ε, διακρίσεις και στους ΛΟΑΔ και στους ανθρώπους με αναπηρία και ειδικά όταν αυτοί ανήκουν στην κοινότητα Ρωμά. Χρειαζόμαστε λοιπόν ισότιμη πρόσβαση ε, στις υπηρεσίες, ε, στις πληροφορίες και χρειάζεται και η υπερχρεωτική εκπαίδευση των θεσμών έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις. Επίσης χρειάζομαστε επιτροπές εθνικής συμφιλίωσης και επιτροπές αλήθειας έτσι ώστε ε, κάποιες διακρίσεις και κάποιες χρόνιες διακρίσεις να περάσουν από αυτές. Δυστυχώς δεν έχουν γίνει αυτά αρκετά σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο έτσι ώστε να παρακολουθούν όλα τα προγράμματα, είτε τα βασικά είτε τα ειδικά για τις μειονότητες και να είμαστε σίγουροι ότι όλη η νομοθεσία εφαρμόζεται με τον σωστότερο τρόπο. Θα δώσω τώρα στον τελευταίο όμως ομιλητή ε, το λόγο που είναι ο κύριος Λος Λαμπουκόφσκι που είναι και ο ε, ε, πληρεξούσης της κυβέρνησης για τις εθνικές μειονότητες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, Καταρχά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αναφέρατε κύριε Πρόεδρε ότι είμαι Σλοβάκος. Αλλά, ε, και γι τον, αλλά θα χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα που είναι τα Ουγγρικά. Αυτό νομίζω ότι εκφράζει ακριβώς ε, πόσο σημαντική είναι η ε, εξασφάλιση της ε, γλωσσικής πολυμορφίας, της πολυγλωσσίας και θέλουμε να σας αναφέρουμε τι δυνατότητες ε, υπάρχουν μέσω του Διεθνούς Νομικού Πλαισίου για την προστασία των μειονοτήτων. Είναι πολύ ευραία τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Μεταξύ αυτών η διασφάλιση των γλωσσικών δικαιωμάτων είναι πολύ βασικό θέμα. Η γλώσσα είναι μέσο επικοινωνίας και είναι, ένα πολύ είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας ενός ατόμου. Έχουν λοιπόν τα γλωσσικά δικαιώματα μεγάλη σημασία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των μειονοτήτων. Αλλά η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βοήθησε σημαντικά τις μειονότητες. Στη δεκαετία του 90 αποφασίστηκαν δύο, δύο διεθνείς συμβάσεις που αναφέρθηκαν και προηγουμένως ε, η χάρτα για την χρήση των περιφερειακών γλωσσών και η σύμβαση πλαίσιο για τα δικαιώματα των μηνοτήτων. Όλα αυτά βέβαια ε, είχαν να κάνουν και με τις ε, φρικτές ε, συγκρούσεις που ξεκίνησαν στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Από εκεί εξήχθησαν ορισμένα πολιτικά πορίσματα ότι πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώματα των μειονοτήτων για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις. Αυτά τα δύο κείμενα για την προστασία των μηνοτήτων καθορίζουν το γενικό πλαίσιο δράσης των κρατών μελών, τα οποία βεβαίως έχουν και αυτά ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν. Το μεγάλο θέμα είναι εάν ε, οι ελπίδες που είχαν δημιουργηθεί μέσω αυτών των δύο συμβάσεων έγιναν πραγματικότητα, εάν δηλαδή υπάρχει ουσιώδης ε, προστασία των μηνοτήτων. Όπως ξέρετε, ε, η χάρτα άρχισε να ισχύει το 1998. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πάνω από 80 περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες. Και πρέπει να πούμε ότι πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν επικυρώσει ή δεν έχουν καν ε, ενταχθεί σε, αυτήν, σε αυτές τις συμβάσεις. Πρέπει όμως πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε τι εννοούμε γλωσσικά δικαιώματα μπορούν να αναγνωριστούν ε, μεμονωμένα ή λειτουργούν μόνο σε σύνδεση με άλλα δικαιώματα. Εγώ θεωρώ, και δεν είμαι ο μόνος, ότι τα γλωσσικά δικαιώματα συνδέονται άμεσα με πολλά άλλα δικαιώματα. Το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης, ελευθερίας της συνείδησης, ε, της θρησκευτική πίστης. Οπότε, η ύπαρξη τελικά των γλωσσικών δικαιωμάτων έχει να κάνει με την ύπαρξη της δημοκρατίας και αντίστροφα. Είναι λοιπόν βασικός πυλώνας της δημοκρατίας τα γλωσσικά δικαιώματα. Παίζουν σημαντικό ρόλο και πρέπει να είναι πάντα εγγυημένα γιατί είναι αναγκαία για να ασκήσουν πολλά άλλα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Το δικαίωμα να εκφράζεται κανείς τη γλώσσα του είναι θεμελιώδες δικαίωμα και είναι μεταξύ των βασικών δικαιωμάτων της δεύτερης και τρίτης γενιάς. Το δικαίωμα αυτό αυτή τη στιγμή προτάσεται ιδιαίτερα και το βασικό είναι να μπορεί κανείς να μιλάει στη γλώσσα του όχι μόνο στον ιδιωτικό βίο αλλά και στην επικοινωνία με τη διοίκηση, στο δημόσιο βίο γενικά στην καθημερινή του ζωή στον κοινωνικό τομέα, στον πολιτιστικό τομέα Όσον αφορά τώρα τον τρόπο ε, έκφρασης αυτών των γλωσσικών δικαιωμάτων πρέπει να υπάρχει και οπτική διγλωσία και πολυγλωσία και να είναι νομικά εγγυημένη. Και πρέπει να καλύπτει ε, το πλήρες φάσμα του ιδιωτικού και δημοσίου βίου. Όμως, το θέμα είναι αν αυτό ε, ισχύει στην πραγματικότητα. Με τι μορφή και σε τι βαθμό. Δηλαδή ε, είναι σαφής και ορατή η δυνατότητα ε, να εκφράζεται κανείς και στη γλώσσα του κράτους και στη γλώσσα της μειονότητας στην οποία ανήκει. Και εδώ παίζουν ρόλο πολλοί κοινωνικοί παράγοντες. Το να μπορεί να το κάνει κανείς αυτό ε, στέλνει σημαντικό μήνυμα. Πρώτα απ' όλα στην ίδια τη μειονότητα που αποκτά αυτοπεποίθηση. Αλλά και η πλειονότητα που δεν ανήκει σε αυτή τη μειονότητα με αυτόν τον τρόπο καταδεικνύει την αποδοχή της και τη δημοκρατικότητά της. Και έτσι ε, στην ουσία προωθείται η κοινωνική ισότητα. Για παράδειγμα το Ρωμά. Να είναι λοιπόν ορατά τα γλωσσικά δικαιώματα με τον κατάλληλο τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει λοιπόν να βασίζεται ε, σε ένα σωστό νομικό πλαίσιο. και πρέπει να υπάρξουν δεσμευτικά νομικά κείμενα και κατόπιν πρέπει να υπάρχει και αναγκαία βεβαίω υποδομή. Πρέπει να υπάρξει η αναγκαία εναρμόνιση των ε, προδιαγραφών αυτών σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό όμω αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Γιατί αυτή τη στιγμή ακόμη τα κράτη-μέλη δεν έχουν εφαρμόσει αυτά που προβλέπουν οι δύο συμβάσει τι οποίε προαναφέρθηκα. Πολλά κράτη-μέλη βεβαίω έχουν υιοθετήσει νομοθετήματα, αλλά στην πράξη υπάρχουν ακόμη πολλά εμπόδια. Σε πολλά κράτη-μέλη πολλές φορές ε, θεωρείται χαρτί στο πολιτικό παιχνίδι η αποδοχή των ε, δικαιωμάτων των μειονοτήτων και λέγεται ότι είναι γενικά θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πολιτών και θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή ε, ρύθμιση των ελαχίστων δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα νομικό δεσμευτικό πλαίσιο. Υπάρχουν όπως σας είπα πολλά προβλήματα. Όμως παρόλα αυτά αυτές οι δύο συμβάσεις είναι σημαντικά μέσα, παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω λοιπόν ότι είναι κατάλληλη συγκυρία για να προχωρήσουμε περισσότερο. Να διευκολυνθεί η αποδοχή ελαχίστων προδιαγραφών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τελική ομιλήτρια, πριν πάρουν το λόγο και οι συνάδελφοι, για να έχουμε μια άλλη προοπτική για τις ε, μειονοτικέ και περιφερειακές γλώσσες είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ε, ημερησιών εφημερίδων στις γλώσσες αυτές ε, η κυρία Σλέζα από την Ιταλία. Ευχαριστώ. Χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα που μπορώ και εγώ να μιλήσω για τις ε, μειονοτικέ και περιφερειακές γλώσσες. Η οργάνωσή μου δημιουργήθηκε πριν από 17 χρόνια με την πρόταση ε, διευθυντών τέτοιων εφημερίδων για να συντονίσουν την ε, ε, δράση για την πληροφόρηση αλλά και για να αποτελέσουν πλατφόρμα για την προώθηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Όπως ξέρετε το αναγνωστικό κοινό αυτών των εφημερίδων είναι πολύ περιορισμένο, άρα δεν υπάρχει πάντα επαρκής χρηματοδότηση και εργάζονται με πολύ, πολύ λίγους ε, συνεργάτες. Έχουμε 27 τέτοιες εφημερίδες που ανήκουν ε, στην Ένωσή μας και έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εμείς ε, τις σημερινές τάσεις της ψηφιοποίησης κτλ. Ορισμένες εφημερίδες χρειάστηκε να σταματήσουν να εκδίδονται, άλλες ε, επολύθησαν σε, μεγάλα, ε, σε μεγάλους ομίλους, σε μεγάλους εκδοτικούς ομίλους. Στην ε, Γαλλικία υπήρξαν εξελίξεις, όπως και στην Σλοβακία, όπου η μόνη εφημερίδα αγοράστηκε από ένα μεγάλο όμιλο. Στην Ισπανία δύο καταλανικές εφημερίδες συγχωνεύτηκαν και αυτό συνέβη και με δύο σουδικές εφημερίδες στη Φιλανδία. Χαιρετίζουμε λοιπόν αυτήν την ε, έκθεση γιατί προωθούμε ακριβώς την ε, πολυγλωσία. Η ενημέρωση των μηνοτήτων στη γλώσσα τους είναι πολύ σημαντική για την εγγύηση της πολιτιστικής του ταυτότητα, ταυτότητας, αλλά και για τη δυνατότητα να εκφραστεί ε, ελεύθερη άποψή τους. Οι μειονότητες μπορεί πολύ εύκολα να είναι σε θέση. Γι' αυτό πρέπει να βοηθήσουμε να υπάρξει ισότητα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι υποχρεωμένα και πολιτικά και νομικά να δημιουργούν το κατάλληλο πλαίσιο που να επιτρέπει να υπάρχει αυτή η πολυγλωσία στα ΜΜΕ. Υπάρχουν εδώ και δεκαετίες αυτές οι ημερήσεις εφημερίδες. Είναι πολύ δεμένες με τη ζωή των μηνοτήτων, έχουν μεγάλη πείρα, γνωρίζουν την κατάσταση των μειονοτήτων. Άρα δεν μας ενημερώνουν μόνο για τη σημερινή πραγματικότητα, αλλά έχουν και μια ιστορική διάσταση. Και ξέρουμε ότι για ε, ορισμένα άτομα σε αυτές τις μειονότητες είναι η μόνη πηγή ενημέρωσης. Και δεν είναι μόνο πηγή ενημέρωσης, αλλά, όπως είπα, μπορούν να είναι και πλατφόρμα για να εκφραστούν αυτές οι μειονότητες, να περάσουν οι απόψεις τους ε, στα εθνικά μέσα. Γιατί δύσκολα ακούγεται τη φωνή των μειονοτήτων στα εθνικά μέσα. Έτσι βοηθάει ε, η λειτουργία αυτών των εφημερίδων τα εθνικά μέσα να ενημερώνουν για την πραγματική κατάσταση των μειονοτήτων και έτσι αποφεύγεται στις εθνικές, ε, στα εθνικά μέσα να υπάρχουν μόνο αρνητικές ιστορίες για τις μειονότητες. Αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση. Σε πολλές ε, χώρες είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητές μας και πολύ περιορισμένες δυνατότητες να λάβουν εθνικές ενισχύσεις. Αυτό αφορά τα έντυπα μέσα, ε, πολύ συγκεκριμένα, που κάνει την κατάστασή τους πολύ δυσχερή, γιατί ούτως ή άλλως είναι δυσχερής από τη φύση της. Και όπως σας είπα, είναι περιορισμένο και το αναγνωστικό κοινό. Οπότε δεν είναι κερδοφόρες αυτές οι επιχειρήσεις. Η δημογραφική δομή αυτών των ε, μειονοτήτων επίσης μας δημιουργεί δυσχέρειες. Γιατί είναι σε μεγάλο βαθμό ηλικιωμένα τα μέλη των μειονοτήτων, άρα δεν έχουν πολλά μέσα και για να αγοράζουν εφημερίδες. και ε, γνωρίζετε ότι η οργάνωσή μας κάνει τη δουλειά που βοηθάει, μας βοηθάει να οργανωθούμε καλύτερα, μπορούμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες και... Πράγματι, το Μίδας μας έχει περίπου 3 εκατομμύρια αναγνώστες. Συμφωνούμε λοιπόν, υποστηρίζουμε την ε, διαδικτυακή την δικτυακή δημιουργία αυτών των ε, ε, τωρινών εντύπων, αλλά θα πρέπει να εγγυηθούμε και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, για να μείνουμε μέσα σε αυτήν την υπόθεση, υπάρχει μία ε, ε, υποτροφία που εγγυάται τις σπουδές σε κάποιους ανθρώπους. Θα πρέπει αυτό να το εγγυηθούμε και για ε, τα ηλεκτρονικά μέσα. Θα πρέπει δηλαδή να προσφέρονται δυνατότητες ε, και υπάρχουν ανάγκες δηλαδή για άλλους, άλλους πόρους χρηματοδότησης για την ε, κατάρτιση των δημοσιογράφων που εργάζονται στα ηλεκτρονικά μέσα για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ανταγωνιστικότητά τους μέσα στο πλαίσιο τέτοιων ειδών εκπαίδευσης θα μπορούσαν μπορούσαμε να μιλήσουμε για την ανοχή, ε, την πολιτιστική, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ε, στο πλαίσιο της δημοσιογραφίας. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση δε, αυτά τα περιοδικά, οι καθημερινές εφημερίδες για τις μηνότητες είναι πολύ σημαντικά μέσα ενημέρωσης γιατί εν γέννη οι μειονότητες έχουν πολύ θετική στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς αυτή θεωρείται δυνατότητα και εγγύηση κοινή και γι' αυτό το λόγο συχνά στα περιοδικά αυτά των μειονοτήτων, στις εφημερίδες των μειονοτήτων τα ευρωπαϊκά ζητήματα βρίσκουν πολύ περισσότερο χώρο από ότι τα ευρέως διαδεδομένα μέσα. Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό να ε, εγγυηθούμε ότι τα μέλη των μειονοτήτων θα είναι παρόντα ως ε, δημοσιογράφοι στην σύνταξη των μέσων ε, των μεγάλων εφημερίδων και στις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και στα όργανα που λαμβάνουν τις αποφάσεις που αφορούν τα έντυπα ώστε να ακούγονται και οι δικές μας φωνές. Πρέπει επίσης να δημιουργηθούν επιτροπές εποπτείας που να μπορέσουν να είναι ένα όργανο προσφυγής και να επιβάλλουν και κυρώσεις σε περιπτώσεις παρατυπιών. Δεν μπορούμε παρά να μιλήσουμε εδώ και για τις νέες τεχνολογίες. Το ίντερνετ είναι πάρα, σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό και για τις μειονότητες βεβαίως. Ωστόσο λείπουν πόροι. Λείπουν δημόσια κονδύλια για να μπορέσουμε να έχουμε εγγυημένη δυνατότητα διάδοσης αυτών των πληροφοριών και βλέπουμε ότι η τεχνολογική ανάπτυξη τόσο στον έντυπο τύπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο προσφέρει τεράστιες δυνατότητες. Για παράδειγμα, αν σκεφτούμε το software μετάφρασης που χρησιμοποιείται στη, στην, στην, ε, όσον αφορά τη μετάφραση των ε, ε, ισπανικών και καταλανικών εντύπων. Όλη αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τις μειονότητες. Χρειάζεται δηλαδή να υπάρξει ειδική κατάρτιση ώστε να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχει τέτοιο είδους προσφορά μετάφρασης μέσω των τεχνολογιών και αυτό πρέπει να γίνει για όλες τις γλώσσες, όχι μόνο για τις επίσημες γλώσσες των χωρών μελών αλλά και για τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες τα γραφεία ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προσέξουν όλος ιδιαίτερο τα μέσα των εθνικών μειονοτήτων. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και εγώ σας. Σε ευχαριστώ όλους τους ομιλητές μας και θα ε, ζητήσω από τον εισηγητή μας να κάνει κάποιες ε, ε, τελικές παρατηρήσεις στο τέλος γιατί όπως οι συνάδελφοι θα έχουν διαπιστώσει, είναι ένα πολύ σπουδαίο ζήτημα το θέμα των μειονοτήτων εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορούμε αυτό να το δούμε και από τις ε, παρουσιάσεις της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Είναι ευρύτατο το θέμα και έχουμε κάνει και άλλες εκθέσεις ε, στην Επιτροπή μας ε, σχετικά. Θα ζητήσω λοιπόν τον κύριο Νάγκη να, να βγάλει τα συμπεράσματά του στο τέλος. Η έκθεση αυτή αφορά κυρίως τις γλώσσες των μειονοτήτων. Το αναφέρω αυτό γιατί στη συζήτηση που κάνουμε σήμερα ε, βασίζεται ε, στις ομιλίες των ομιλητών που καλέσαμε για αυτό το θέμα, αλλά μιλήσατε και για άλλα θέματα, γιατί υπάρχουν και άλλες εκθέσεις που θα συνταχθούν για ένα σωρό ζητήματα που αφορούν τις μειονότητες. Αυτή είναι η τελευταία. Το αναφέρω για να σας δώσω το πλαίσιο. Ο κύριος Σόγκορ πρώτα. Πόση ώρα έχω. Ένα λεπτό. Άντε και δύο, αν θέλετε. Θα μιλήσω με, χρησιμοποιώντας μόνο τα, κυριότερα ζητήματα. Το θέμα του ορισμού των μειονοτήτων είναι πολύ σημαντικό το και επανέρχεται. Νομίζω θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στις ευθύνες των κρατών μελών ή μάλλον να πω την ανευθυνότητα των κρατών μελών σε σχέση με τις ε, οδηγία κατά των διακρίσεων. Δεύτερον, η εφαρμογή. Σήμερα μιλάμε περισσότερο για την μη εφαρμογή καθώς πρόκειται για μια συστηματική μη εφαρμογή αποφάσεων ε, ε, ρυθμίσεων και κανόνων που δεν εφαρμόζονται και στη χώρα μου, τη Ρουμανία, ε, ε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς οι διαδοχικές κυβερνήσεις ε, αντιμετωπίζουν τη, ως προαιρετική την εφαρμογή των διοικητικών τους αυτών καθηκόντων όσον αφορά την επανεθνικοποίηση της, των εκκλησιών, των μειονοτήτων, ανέχονται το κηρύγματα μίσους και, και ούτω καθεξής Κάποιος ανέφερε τις περιορισμένες αρμοδιότητες σε σχέση με τη, της Ευρωπαϊκής Καλύτερα είναι να εστιάσουμε όμως την προσοχή μας στις δυνατότητες και όχι στους περιορισμούς. Τα, τα, θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να γίνονται σεβαστά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο αν υπάρχει ένα σύστημα προστασίας των μειονοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση με υψηλά προδιαγραφές και υποπτία. Μόνο η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μπορεί να επιβάλλει αυτά τα δικαιώματα. Το Ευρωκοινοβούλιο ήδη έχει ζητήσει τέτοιο είδου ε, σύστημα προστασίας ε, σε αυτή την ε, θητεία και στηρίζει το μηχανισμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την έκθεση, μέσα στην έκθεση μάλιστα για τα, την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια μιλήσαμε επίση για αυτό το θέμα. Τι χρειάζεται για να μπορέσουμε επιτέλους να κινήσουμε αυτό το θέμα. Ο κύριος Γιούρακ, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές και να σας πω το εξής. Ε, ποιο είναι το δικαίωμα για τη συλλογική μνήμη. Ποιο είναι το δικαίωμα που επιτρέπει τη χρήση της μητρικής γλώσσας. Δικαιώματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ε, ταυτότητα καθενός από μας. Οπότε πιστεύω ότι πάρα πολλά από τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στην Ευρώπη ε, ξεσπάνε επειδή ακριβώς δεν έχουμε τις κατάλληλες πολιτικές και επειδή δείχνουν αδράνεια οι θεσμοί οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν την αρμοδιότητα για την προώθηση των δικαιωμάτων μειονοτήτων. Επίσης, η δράση της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς έχουμε απευθύνει εκκλήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλές φορές και η απόκριση που μας δόθηκε ήταν πως το θέμα αυτό δεν αποτελεί δική μας αρμοδιότητα. Και γι' αυτό πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τον Πρόεδρο, όπως επίσης και όλους όσους συμμετείχαν σήμερα στην ακρόαση γιατί με ιδιαίτερη ικανοποίηση είδα πως μπορούμε τουλάχιστον να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Για παράδειγμα, έχουμε προβλήματα με τη μεγαλύτερη γειτονική μας χώρα που είναι η Γερμανία. Εδώ και 30 χρόνια ισχύει μια διμερή συμφωνία με τη χώρα αυτά και έχουμε μια υποχρέωση η οποία είναι η εξής. Θα πρέπει να εξασφαλίζουμε το δικαίωμα ε, στην παιδεία ε, που θα υποστηρίζει την εθνική ταυτότητα. Ωραία όλα αυτά, αλλά έχουμε τα προβλήματα που δημιουργούν το Judentamt στη Γερμανία, το οποίο σημαίνει ότι πολλά παιδιά δεν μπορούν να μιλούν πολωνικά με τους γονείς τους και κάθε προσπάθεια που έχουμε κάνει που είναι να αντιδράσουμε ε, στην επιβολή αυτής της ε, του Ιδρύματος για τους Νέους ε, δεν έχουν δώσει καρπό γιατί δεν έχουμε καταφέρει ε, να επιβάλλουμε το σεβασμό αυτών των διατάξεων. Και το πρόβλημα με το Ίδρυμα αυτό για τη νεολαία και τους νέους είναι πως δεν κάνει καμία προσπάθεια και δεν δείχνει καμία κατανόηση για το γεγονός πως έχουν δικαίωμα τα παιδιά να μιλάνε τη μητρική τους γλώσσα με τους, με τους γονείς τους και πως αυτό είναι ουσιαστικό και πως δεν μιλάμε για μια γλώσσα η οποία ε, χρησιμοποιείται σε μια απόσταση ε, εκατοντάδων ε, χιλιάδων χιλιόμετρων από τα σύνορα της Γερμανίας όχι, είναι μια ε, γειτονική γλώσσα, ε, μια γλώσσα μητρική για ε, ανθρώπους που βραβεύτηκαν με το βρεβείο Νόμπελ και δείχνουν να αγνοούν μια βασική ανθρώπινη ελευθερία. Εδώ προσπαθούμε εμείς να δώσουμε μια μάχη και σας ευχαριστώ για μια φορά ακόμα που φέρνετε το θέμα αυτό στην επιφάνεια και που προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το θάρρος που δείξατε και για το θάρρος με τον οποίο στην έκθεσή σας βάζετε κάποιες ερωτήσεις. Ο κύριος Βελέρο, επόμενος ομιλητής. Thank you very much. Κυρία Βελέρο, με συγχωρείτε, σας ευχαριστώ πολύ. Αν ξεκινήσουμε από την αφετηρία θα δούμε ότι υπάρχουν και ευρωπαϊκές συμβάσεις και η διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε επίσης και την συμφωνία, τη σύμβαση πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και σε όλες αυτές τις συμβάσεις έχουμε κάποιες διατάξεις, οι οποίες είναι υποχρεωτικέ, αλλά είναι υποχρεωτικέ δεσμευτικέ σε διακρατικό επίπεδο. Δεν είναι δεσμευτικέ για τον ίδιο τον πολίτη. Και βέβαια έχουμε και τη δική μα ε, ε, συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 2, που νομίζω θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική για τα ευρωπαϊκά ε, για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς όμως σε επίπεδο δευτερογενούς δικαίου δεν βλέπω να υπάρχει κάτι ικανοποιητικό και βρισκόμαστε στην εξή κατάσταση οι μειονότητε να αντιμετωπίζουν πολύ άσχημη μεταχείριση στην Ευρώπη και αναφέρομαι κυρίως στους πληθυσμούς Ρωμά. Νομίζω λοιπόν ότι όντω έχουμε πρόβλημα μεγάλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν επιβάλλουμε κάποια ελάχιστα πρότυπα ή προδιαγραφέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει τουλάχιστον αυτό να γίνει μέσω κάποιου μηχανισμού ε, που θα τα καταφέρει στην πράξη. Γιατί ο τρόπο με τον οποίο γίνεται σήμερα είναι ο εξή. Το κράτο μέλο καλείται να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των πολιτών του και δεν μπορούμε εμεί να κάνουμε τίποτα. Και βλέπουμε τι γίνεται σε πολλά σημεία τη Ευρώπη. Δεν είναι μόνο τα δικαιώματα των μειονοτήτων που αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν είναι και ε, τα δικαιώματα άλλων κατηγοριών πολιτών και εμεί δεν κάνουμε τίποτα. Πού θα βρούμε λοιπόν μια λύση και ποια θα είναι η λύση αυτή, με ποιο τρόπο μπορούμε εμεί πράγματι να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη σέβονται τι υποχρεώσει του. Χρειάζεται κάποιο είδο μηχανισμό και θα ήθελα να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι είδο μηχανισμό θα ήταν αυτό, τι χρειαζόμαστε άραγε. Εξαιρετική παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ και απευθύνω την ερώτηση αυτή, μια και μα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αρμοδιότητα, μια και έχουμε τις οδηγίες τώρα για ε, κατά των ε, διακρίσεων και αυτό αποτελεί δική μας ε, αρμοδιότητα πλέον και όχι μόνο αρμοδιότητα που μοιραζόμαστε με την Επιτροπή απασχόληση. Λοιπόν, οι οδηγίες αυτές ήταν αρκετά ε, γενικές, αλλά θέλω να μου πείτε τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε τις μειονότητες, πώς θα το ορίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Τροπή. Πολύ καλά αυτά που έχει πετύχει μέχρι σήμερα, αλλά πώς θα τα επιβάλλουμε, γιατί νομίζω ότι υπάρχει πολιτισμικό και νομικό πρόβλημα εδώ. Το τονίζω για να μην ξεχαστεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ο κύριος Φράντς είναι ο επόμενος μιλητής. Σας καλωσορίζω. Νομίζω σας καλωσόρισα και στην τελευταία συνεδρίαση. Δεν φορούσα τα ακουστικά. Είστε νέο μέλος στην Επιτροπή μας και θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Ευχαριστώ πολύ. Εάν δεν ξέρουμε ότι οι Ρώμα δεν λαμβάνονται υπόψη για το καθορισμό της τραγικής στρατηγικής για την ε, συμπερίληψή τους. Και από την πείρα μας ξέρουμε ότι αν δεν γίνεται κάτι τέτοιο δεν έχουμε καμία πιθανότητα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το να γίνεται ταμπού ε, οποιαδήποτε κριτική κατά τον Ρωμά δεν βοηθάει. Και το να μαθαίνουν την ε, ε γλώσσα της χώρας τα γερμανικά, τα γερμανικά συγκεκριμένα δεν βοηθάει εάν δεν συμμετέχουν στα κανονικά σχολεία και αν δεν έχουν τη διάθεση να συμμετάσχουν στην κοινωνία. Η βάση για μια σωστή αντιμετώπιση στην εκπαίδευση δεν έχει προχωρήσει, σχεδόν δεν υπάρχει στην Ανατολική Ευρώπη. Ο αποκλεισμό είναι ο κανόνας για τους Ρωμά, ιδιαίτερα για τα παιδιά τους. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών και για την ε, Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να εφαρμοστεί. Δυστυχώς στη χώρα μου, στη Γερμανία, αυτά τα δικαιώματα ε, παραβιάζονται και όποιος τα παραβιάζει δεν τιμωρείται. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι η διαφθορά που για παράδειγμα δεν επιτρέπει οι πιστώσεις ε, που δίδονται για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά να πάνε πραγματικά σε αυτούς. Πρέπει οι μη κυβερνικές οργανώσεις να συμπεριληφθούν αν θέλουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Γι' αυτό Πρέπει να υπάρξουν και αναγκαίες δομές. Αυτό πρέπει να το προωθήσουμε, να έχουν τις δικές τους δομές. Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Εάν οι αφορόμενοι πρέπει όχι απλώς να καλούμε να συμμετάσχουν, αλλά να, συμμετέχουν και στην πράξη. Ο αντιαθηγανισμός είναι ε, εξίσου καταδικαστέ όσο και αντισημιτισμός. Εδώ και αιώνε ζουν μεταξύ μα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άντεμα. Ευχαριστώ πολύ. Η διατύπωση ελαχίστων προδιαγραφών προστασίας των μειονοτήτων στην Ένωση είναι πολύ σημαντικό θέμα όπως είπε ο κύριος Νάγκη, έχουμε 50 εκατομμύρια πολίτες στην Ένωση που ε, εντάσσονται στα κριτήρια για να αποτελούν μέλη εθνικών μενοτήτων. Αλλά βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν πολύ διαφορετικές στάσεις. Δεν υπάρχει αναγκαία αποδοχή, η αναγκαία καλή θέληση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει όντως να θέσει το θέμα της προστασίας των μειονοτήτων ως προτεραιότητα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξουν ευρωπαϊκά, πανευρωπαϊκά μέτρα και προδιαγραφές για να γίνονται σεβαστά όλα τα άτομα που συμμετέχουν που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες που έχουν συγκεκριμένες ανάγκες. Πρέπει να υπάρξει πλήρης οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ισότητα σε όλους τους τομείς της ζωής. Άρα πρέπει να έχουμε τις αναγκαίες προδιαγραφές για να τις προστατεύουμε. Και πρέπει να ε, ισχύσουν και, για τις, ε, τα κράτη-μέλη και για τις υποψήφιε χώρες, ιδίως τα Δυτικά Βαλκάνια. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θέλει κανένα άλλος συνάδελφος να πάρει το λόγο. Α, βλέπω κύριε Νάγκη, μόλις καθίσατε Θέλετε να κάνετε μερικές καταληκτικές παρατηρήσεις. Νομίζω ότι όσοι συνάδελφοι έχουν ασχοληθεί με τα θέματα των μειονοτήτων ε, τα τελευταία χρόνια από την Επιτροπή μας έχουν ασχοληθεί με διαφορετικές πλευρές. Είναι πολύ ευρύ το θέμα. Έχει να κάνει με φιλετικές και εθνικές μειονότητες, γλωσσικές μειονότητες, καταπολέμηση των διακρίσεων και εγώ έκανα μια έκθεση το 2004 αμέσως μετά την ένταξη κάποιων χωρών Προσπαθούμε λοιπόν να καλύψουμε όλες τις πλευρές εντός των ε, νομικών πλαισίων που έχουμε. Το ανέφερε η κυρία Βαλέρο. Είναι πολύ περίπλοκο και ευρύ το θέμα. Ο εισηγητής βέβαια ασχολείται με μια συγκεκριμένη πλευρά του και ελπίζω ότι μέσω της ακροάσεως καλύψαμε και ορισμένες άλλες πλευρές που δεν είναι απλώς ε, αρμοδιότητα της Επιτροπής μας αλλά και μας ενδιαφέρουν. Κύριε Νάγκη, Θέλετε να κάνετε κάποιες κατακριτικές παρατηρήσεις για το τι θέλετε να επιτύχετε μέσω της εκθέσεώς σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές, λοιπόν, για τα όσα είπαν και κυρίως τον κύριο Μπουκόφσκι, που είναι ο πληρεξούσιος για τις εθνικές μειονότητες από τη Σλοβακία, ο οποίος ουσιαστικά ε, εξέφρασε πολλά από τα όσα θα είχα πει εγώ που έχουν να κάνουν και με μια αντίδραση στο είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη-μέλη. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη όλα τα σχετικά ψηφίσματα, τα εξαιρετικά ψηφίσματα που έχουν ε, ληφθεί στο παρελθόν. Ο κύριος Λέντικερ μίλησε για τα όσα έχουν συμβεί από το 1949 ε, που αναφερθήκαμε ε, στις διατάξεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων είναι ένα διεθνές νομικό εργαλείο το οποίο είναι δεσμευτικό και το οποίο προστατεύει τα δικαιώματα αυτών το οποίο έχει επικυρωθεί από τα 24 από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δυστυχώς όπως είπαν και οι συνάδελφοι το θέμα είναι η εφαρμογή αυτών των διατάξεων από τα κράτη-μέλη όχι μόνο η επικύρωση. Το Συμβούλιο της Ευρώπης παρακολουθεί δραστήρια τα θέματα αυτά και πάρα πολλές καταγγελίες ε, καταφθάνουν συνέχεια και στην τελευταία έκθεση για τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνουμε ότι έχουμε πάρα πολλές παραβιάσεις αυτών των δικαιωμάτων από τα κράτη-μέλη, ακόμα και κάποια βασικά μειονοτικά δικαιώματα. Ξέρετε κι εσείς πως υπάρχει βέβαια ο χρυσός κανόνας, αλλά δεν είναι πάντα απόλυτα δεσμευτικά αυτά και γι' αυτό έχουμε και τα κριτήρια της Κοπεχάγης για τα υποψήφια κράτη προς ένταξη. Νομίζω πως αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε 50 εκατομμύρια πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκουν σε μειονότητες και που απαιτούν να ε, δημιουργήσουμε τα εχέγγυα που θα εξασφαλίσουν το σεβασμό των ε, ε, δικαιωμάτων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είδατε πως μαζέψαμε και 1,4 εκατομμύρια ε, υπογραφές στο σχετικό ε, θέμα. Έχουμε και την απόφαση του ΔΕΚ για την πρωτοβουλία αυτή της εθνικής μειονότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, όπως είπε και η δική μας έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα, χρειαζόμαστε ελάχιστα πρότυπα για τις εθνικές μειονότητες και για τις εθνοτικές ομάδες γνωρίζουμε ποια είναι τα όρια των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντω σε άλλε πολιτικέ είναι πάρα πολύ ευέλικτη στο θέμα αυτό και θεωρώ πω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την ευθύνη ε, στο να προωθεί τα θέματα αυτά, στο να σπρώχνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να βρει αυτό το περιθώριο ε, για να δώσει κάποια απόκριση και να ε, υποχρεώσει ε, τα κράτη-μέλη τα οποία δεν σέβονται αυτόν τον χρυσό κανόνα. Και εσείς, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τι πιστεύετε για το ΔΕΚ. Γιατί δεν είναι μόνο το 1,4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες που υπέγραψαν ε, σε αυτή την εκστρατεία που έγινε, αλλά είναι και το ΔΕΚ σας υπενθυμίζω. Εσείς αυτό πώς το αντιμετωπίζετε. Θέλετε να αποφασίσετε, να απαντήσετε τώρα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, θέλω να διευκρινίσω κάτι για την απόφαση ε, του Γενικού Δικαστηρίου, πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε αυτό το πακέτο για την μειονότητα ε, βάσει κάποιων κριτηρίων. Είναι 11 προτάσεις για νομική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρχικά την απορρίψαμε γιατί δεν μπορούσε να παρουσιάσει ένα πλήρες πακέτο προτάσεων και για τα 11 αυτά θέματα. Το δικαστήριο λοιπόν αποφάσισε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει εξειδικευμένα να αντιμετωπίσει κάθε μία από τις 11 προτάσεις, να τις μελετήσει, το κάναμε και εγκρίναμε μόνο δύο από τις 11, οι οποίες, ε, ε, συγγνώμη, είπαμε ότι μόνο δύο από τις 11 είναι εκτός αρμοδιότητας, άρα λοιπόν εγκρίναμε μερικό στο πακέτο και όταν ε, υποβληθούν για αυτά τα νέα, νέα θέματα θα πρέπει μέσα στους τρεις μήνες να δώσουμε μια απάντηση αλλά για το κατά πόσο έχουμε γενικότερη αρμοδιότητα για τα ελάχιστα πρότυπα για τις εθνικές μειονότητες, όχι. Δεν ε, ισχύει κάτι τέτοιο. Βεβαίως δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να προδικάσουμε τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρωτοβουλία πολιτών αυτή. Όταν κατατεθεί θα γίνει και ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω πως τα όσα ακούσαμε από τα μέλη μας, στους ευρωβουλευτές, ήταν πολύ καλές ε, προτάσεις και σχόλια για το τι συμβαίνει ε, με τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τους ελάχιστους κανόνες. Είναι ένα ευρύ και ιδιαίτερα περίπλοκο θέμα. Έχουμε και την έκθεσή μας, που είναι η έκθεση Νάγκη, την οποία θα τροποποιήσουμε ε, με τον κατάλληλο τρόπο και σας ευχαριστώ που κάνατε αυτή την ακρόαση έτσι ώστε να συνδυαστεί με τη δική σας έκθεση. Ευχαριστώ συνάδελφοι για τα σχόλιά σας και ιδιαίτερα ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας για τις εξαιρετικές παρεμβάσεις τους. Σας ευχαριστώ λοιπόν για το χρόνο που μας διαθέσατε. Ποτέ δεν φτάνουν τα όσα κάνουμε για, τις, τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Ε, σας ευχαριστώ πάντως. Είναι απόλυτη αρμοδιότητα της Επιτροπής μας και επαναλαμβάνω πως ευχαριστώ και τα μέλη μας που συμμετείχαν στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ όλους. go with the presentation by the Commission and afterwards to give the floor to Mrs. Metzola, who's reading something. From Mrs. Omar. Yes. So, colleagues, um... Συνάδελφοι, όσοι δεν επιθυμείτε να μείνετε για την, συζήτηση, επόμενη συζήτηση, παρακαλώ να είστε ήσυχοι. Επόμενο σημείο είναι η θέσπιση ενός ταμείου για την εσωτερική ασφάλεια. Πρόκειται για την πρόταση που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή για την, για την ε, εσωτερική ασφάλεια ως τμήμα της επόμενης πολιτικής ε, ε, πενταετίας, μέχρι το, μάλλον δεκαετίας μέχρι το, το 27. Η κυρία Χολμάγερ είναι άρρωστη και την αντικαθιστά ο... η Ρομπέρτα. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα την παρουσίαση της ε, Επιτροπής. Έχουμε κάποιο συνάδελφο εδώ από την ε, Γενική Διεύθυνση Home. να περιμένουμε λίγο να φύγουν όσοι συνάδελφοι θέλουν να φύγουν μετά το τέλος της ακρόασης για να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ρομπέρτα, αντικαθιστά στην κυρία Χολμάγερ. Ωραία, λοιπόν. Αν μπορεί ο συνάδελφος από την ε, DG Home να μας πει ποια είναι τα γενικά κύρια χαρακτηριστικά αυτού του ομέσου και μετά θα ζητήσουμε από την κυρία Μετζόλα να δώσει την ε, ε, θέση της εισηγήτρια. Μάλιστα, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε ε, να είμαστε σήμερα εδώ. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, έχουμε ένα νέο ταμείο που έχει το ίδιο Έχουμε λοιπόν το ίδιο ταμείο αλλά με διαφορετικό όνομα, με, μάλλον το ίδιο όνομα με το νέο ε, όρο. Έχουμε προστιθέμενη αξία λοιπόν για τις δράσεις των ε, κρατών μελών. Βλέπουμε κάποια παραδείγματα ποια, ε, για το ποια είναι η προστιθέμενη αξία. Φυσικά, προωθείται, προωθούνται οι εθνικές δυνατότητες, εκπαιδεύονται οι, ε, ε, αρμόδιοι για την επιβολή ε, του νόμου και όλα αυτά έχουν προσθέσει τη αξία στην συλλογική ευρωπαϊκή δράση εντός της Ένωσης. Συμπέρασμα είναι λοιπόν και περνάμε στην επόμενη διαφάνεια ότι το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου είναι το σωστό και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην στο έγγραφο το οποίο έχετε λάβει. Ε, ε, επίσης μάθαμε ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, κάποια προβλήματα το κύριο ήταν η έλλειψη ευελιξίας. Θα δείτε κάτι, θα επανέλθουμε νομίζω όταν θα παρουσιάσουμε το άμυφ, το θέμα δηλαδή για το άσυλο ε, και θα δείτε ότι υπήρχε έλλειψη ευελιξίας που εμπόδιζε την Ένωση να ε, δράσει να ε, χορηγήσει τα κονδύλια στις σωστές προτεραιότητες. Ε, Επίση, χρειάζεται περισσότερη απλοποίηση. Αυτό είναι κάτι που πάντα ε, χρειάζεται, ε, γιατί συνήθω τα ταμεία είναι κάπω περίπλοκα. Έχουμε επιτύχει ένα βαθμό απλοποίηση, αλλά ακόμα προσπαθούμε σε αυτό το τομέα. Τέλο, ένα μεγάλο λάθο που κάναμε, αν θέλετε, στο παρελθόν είναι ότι πολύ αργούσαμε με την κοινή το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης. Πολύ αργούσαμε όσον αφορούσε μια σαφή ιδέα προς τα μέλη πώς και ποιε βάσεις θα πρέπει να αξιολογούν. Τώρα, εδώ, για να δούμε πώς λειτουργεί η καρδιά αυτού του, του, του, του ταμείου. Έχουμε λοιπόν ότι αντίθετα με το παρελθόν, έχουμε ασφάλεια σε ένα διαφορετικό κεφάλαιο από την μετανάστευση και τα σύνορα, μαζί με την άμυνα και την πολιτική προστασία. Υπάρχουν ε, επιχειρήματα υπέρ και κατά, αλλά αυτή είναι η πρότασή μας και πιστεύουμε πως είναι λογική. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δείτε πως το Ταμείο έχει πολλαπλασιαστεί ε, στο, κατά 1,8 εάν περιλάβουμε και τους οργανισμούς. Επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπουμε πιο συγκεκριμένα τον ε, καταμερισμό ε, για τις εσωτερικές υποθέσεις αυτά τα, τα κονδύλια που πάνε στους οργανισμούς αλλά και στο ίδιο το Ταμείο. Θα θυμάστε βέβαια έχουμε τις EPOL, Europol, MCDDA οι υπηρεσίες, οι οργανισμοί για την ασφάλεια χρηματοδοτούνται χωριστά από το Ταμείο Ασφάλειας. Δεν πληρώνει αυτό για τους οργανισμούς. Είναι δύο διαφορετικά κονδύλια. Ε, οι οργανισμοί έχουν τα δικά τους μέσα. Θα δείτε λοιπόν ότι το Ταμείο εσωτερική Ασφάλειας παίρνει το 7% τη συνολικής χρηματοδότησης, έχει πολλαπλασιαστεί επί 2,5% που φέρνει τα ποσά από το 1 ε, εκατομμύριο στα 2,5. Και το Ταμείο για την Ασφάλεια θα λάβει ε, χωριστό ποσό. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε και την περιγραφή, σύντομη περιγραφή του πεδίου εφαρμογής αυτού του ε, Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Θα δείτε ότι αυτό το Ταμείο ε, αφορά οριζόντια θέματα. Πρώτον, υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ιδιαίτερα καταπολέμηση και ε, αντιμετώπιση του τρομοκρατία, ε, τη ριζοσπαστικοποίηση των ε, σοβαρών ε, εγκλημάτων και μιας νέας απειλής που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το κυβερνό έγκλημα. Έχουμε και πιο συγκεκριμένους στόχου που είναι ο πίδη οριζόντι, δηλαδή αύξηση της ανταλλαγή πληροφοριών, που είναι προφανώς ένα από τα προβλήματα ε, στη τομέα της ασφάλειας της Ένωσης, εντοτικοποίηση των διασυνοριακών ε, επιχειρήσεων, ε, και ισχυρότερη δυνατότητα ανθεκτικότητας και αντιμετώπισης των διασυνοριακών εγκλημάτων. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε τους συγκεκριμένους στόχους και τους υποστόχους, δράσεις ή προτεραιότητες. Η ανταλλαγή πληροφοριών λοιπόν, βασικά θα χρηματοδοτήσουμε συστήματα πληροφορικής ε, όπως το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, αλλά βέβαια αλλά όχι μόνο τη δημιουργία συστήματων πληροφορικής αλλά και την ε, πραγματική χρήση πολύ ωραία είναι να έχουμε καλά και ενήμερα συστήματα, μοντέρνα, αλλά πρέπει και ο κόσμος που τα χρησιμοποιεί να είναι εκπαιδευμένος για τα χρησιμοποιήσει, να μπορεί να ανταλλάξει τις πληροφορίες και να τις ερμηνεύσει με εναρμονισμένο τρόπο και ανάμεσα στα κάτι μελη να ανταλλάσσονται πληροφορίε, αλλά και ανάμεσα στου διάφορους αρμόδιου φορείς. Ε, τώρα, εφαρμογή κοινέ ερευνητικέ ομάδες, το γνωρίζουμε ήδη αυτό από το τωρινό ταμείο, κοινέ επιχειρήσεις, πολύ συγκεκριμένε δράσει και στη συνέχεια εφαρμογή δράσεων αντικτύπου που είναι συνήθω οι δράσει που είναι πολύ γνωστές ε, μέσα στο θέμα της, ε, ε, του κύκλου πολιτικής. Ε, τώρα, ενδυνάμωση και συνέχιση δικτύων που έχουμε ήδη φτιάξει, Airpol, Interpol κτλ. Δίκτυα που χρειάζεται να συνεχιστούν. Καθώς και, και ανα, αναβάθμιση. Και βεβαίω να βελτιώσουμε και τι βέλτιστε πρακτικέ και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών επιβολή του νόμου και συνεργασία με τη ΣΕΠΟΛ, την Europol και την MCDDA και άλλου εθνικού φορεί των κρατών μελών. Τρίτος στόχος. Αναλυτικά να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας, να βοηθήσουμε την κατάρτιση, τους διάφορους εμπλεκόμενους, ιδιαίτερα τις ε, αστυνομικές αρχές, τις ε, νομικές υπηρεσίες, αλλά και την κοινωνία ευρύτερα, να ενημερώσουμε, να αυξηθεί η συνειδητοποίηση. αλλά με μία επιφύλαξη. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν πάρει τη μύρδα του λέοντος ε, της χρηματοδότησης. Όμως αυτό δεν έχει αποδειχθεί τελικά ως ε, ο καλύτερος τρόπος ε, προσθήκης ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Ίσως καλύτερα να μην δαπανούμε τόσο πολλά για εξοπλισμό, ιδιαίτερα τον βασικό εξοπλισμό. Αργότερα λοιπόν θα πούμε ότι δεν είναι επιλέξιμες οι βασικές ε, δεν είναι επιλέξιμος ο βασικός εξοπλισμός, για παράδειγμα τα περιπολικά. Αυτά πρέπει να τα πληρώνουν τα κράτη-μέλη και θα το περιορίσουμε στα 15% τους ή άλλους. Και όπως σας είπα, η κατανομή των πόρων, πολύ σημαντική, να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε τους διάφορους οργανισμούς, Europol, Sepol και η e έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά μέχρι τώρα, αυξάνουμε τη χρηματοδότησή του. δεν είναι σαφή ο καταμερισμό ακόμη, θα υπάρξει πιο συγκεκριμένη πρόταση μέσω της ετήσιας διαδικασίας του προπολογισμού. Επίσης θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε οι φορείς αυτοί να συμμετέχουν όχι μόνο στην εφαρμογή, αλλά περισσότερο και στην ε, προγραμματική φάση, για να εργαστούμε χέρι με χέρι με τους οργανισμούς αυτούς για τον προγραμματισμό για το 2021, αλλά και για τη φάση εφαρμογής. Λοιπόν, πώς χρηματοδοτούμε τα κράτη-μέλη. Δεν είναι τα κριτήρια που παρουσιάζω εδώ, αλλά η κατανομή. 2,5 δις είναι ο συνολικός φάκελος. 1,25 δις, τα μισά, θα δίδονται αρχικά, στην αρχή της περίοδου, στα εθνικά προγράμματα των κρατών μελών. Χρειάζεται όμως να υπάρχει μεγάλη ευελιξία Κάνουμε λοιπόν μια κάπως ε, ριζική πρόταση. 50% του υπόλοιπου 50%, δηλαδή 25%, θα πρέπει να δοθεί σε όλη την περίοδο 21-27, 10% κατά τη φάση της ενδιάμεσης αναθεώρησης. Την προηγούμενη φορά δυστυχώς, δυστυχώς για το Κοινοβούλιο, χάσαμε την ευκαιρία να εκταμιευθούν πόροι κατά την αναθεώρηση. Άρα ήταν εξεδοντιασμένη η αναθεώρηση γιατί δεν μπορούσε να αποφασίσει επί της χρηματοδοτήσεω. Ε, επανεξετάσαμε τι προτεραιότητε, αλλά δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε τη χρηματοδότηση. Κρατάμε λοιπόν 250 εκατομμύρια που θα εκταμιευθούν το 2024, θα αποδοθούν. Με τα ίδια κριτήρια με το 2021, αλλά με τις τελευταίες στατιστικές. Θα αποκληθεί η θεματική διευκόλυνση. Κάθε δύο χρόνια θα καθορίζουμε τις προτεραιότητές μας που θα συζητώνται μέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας. Τώρα λοιπόν, να και τα κριτήρια για την απόδοση των πιστώσεων ανακράτος μέλος. Θα είναι τρία πολύ ουδέτερα κριτήρια. 40% ανάλογα με τον αριθμό του πληθυσμού, 15% με βάση την επικράτεια και 45% αντιστρόφως ανάλογα με το ΑΕΠ. Δηλαδή οι φτωχότερες περιοχές θα πάρουν περισσότερα. Είπαμε λοιπόν, 40% έχει να κάνει με το μέγεθος του πληθυσμού και 15% με το μέγεθος της επικράτειας. Σκεφτήκαμε πολύ και για κριτήρια που να έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, γιατί αυτά δεν έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Αλλά μέχρι στιγμή ε, υπήρξε αδύνατο να καθορίσουμε κριτήρια που να ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη, που να είναι αξιόπιστα, που να ε, έχουμε στοιχεία για αυτά τακτικά, για να τα χρησιμοποιήσουμε για την ε, κατανομή των πόρων. Αντί λοιπόν να έχουμε αυτά τα αναξιόπιστα στοιχεία, κρατήσαμε αυτά τα τρία αξιόπιστα βελτίωση της ε, χρηματοδότησης, περισσότερη ευελιξία είναι σχετικά ριζική η πρότασή μας, ριζικά διαφορετική και θα έχουμε και περισσότερες δυνατότητες να υποβάλουμε όρους. Θα έχουμε συγκεκριμένες ε, συστάσεις από τη διαδικασία ε, αποτίμησης του Σέγγεν και Βεβαίω γενικά ήδη αξιοποιούν αυτές τις συστάσεις για να εφαρμόσουν ε, τα κριτήρια, αλλά θα το κάνουμε πιο υποχρεωτικό. Επίσης, άλλη προπόθεση. αν υπάρχει διαδικασία επιπαραβάση για κάποια προτεραιότητα ή δράση, τότε θα αναστέλλονται οι πληρωμές. Άλλη καινοτομία. Κάτι που ήταν πολύ χρήσιμο για τα σύνορα, για το Ταμείο των Συνόρων να ισχύσει και για το Ταμείο αυτό. Θα πληρώνουμε το 100% του λειτουργικού κόστους για τα συστήματα πληροφορικής. Έτσι θα εφαρμοστεί ταχύτερα το Ταμείο. Αλλά θα το περιορίσουμε στο 10%. Και θέλουμε να υπάρχει καλύτερη ευθυγράμμιση με τις νομοθετικές προτεραιότητες και θα αξιοποιήσουμε και ε, συμφωνίες ε, συνεργασίας με τα διαθροτικά ταμεία. Θα αξιοποιήσουμε δηλαδή τη συνεργασία με άλλα ε, στοιχεία του ISF, του Ταμείου Ασφάλειας. Γιατί ξέρουμε ότι είναι περιορισμένοι οι πόροι και ιδίω οι πόροι των διαθροτικών ταμείων. Μια νέα βελτίωση του ταμείου είναι ότι θα υπάρχει υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότηση για συγκεκριμένες δράσεις που θεωρούμε ότι προσφέρουν ιδιαίτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία πολέμηση και πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και διαλειτουργικά συστήματα προφορικής. Κάποιες δράσεις τις θεωρούμε πλέον μη επιλέξιμες. Δηλαδή θέματα που έχουν να κάνουν με στρατιωτική ε, δραστηριότητα ή ε, διαδικασίες ή εξοπλισμός ε, άσκησης βίας. Εδώ σας εξηγώ τι σημαίνει ευελιξία. Υπάρχει η θεματική διευκόλυνση όπως σας είπα και η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Εδώ βλέπετε πώς λειτουργεί η θεματική διευκόλυνση. Αριστερά βλέπετε το 50% των πόρων που θα κατανεμηθούν το 2021. Κατόπιν 10% το 10% που είναι σε αυτό το γκρίζο κουτί που θα αποδοθεί κατά την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση το 2024. Με τα ίδια κριτήρια το 50% αλλά με βάση τα τελευταία στατιστικά στοιχεία των τελευταίων τριών ετών. Το, 20, το 2024 θα έχουμε τα στοιχεία του 2023 διάθεσή μας, ενώ το 2020 θα έχουμε τα στοιχεία του 2019-2020, ανάλογα με τα τελευταία που θα έχουμε. Και από την άλλη πλευρά έχουμε κάποια ευελιξία για τη θεματική διευκόλυνση. Τι είναι η θεματική διευκόλυνση τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τα διάφορα μέσα που ήδη έχουμε, για παράδειγμα επίγουσα βοήθεια, ενωσιακέ συγκεκριμένε δράσει, ούτω ώστε να αποδοθούν πόροι στι προτεραιότητες με υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Γιατί τώρα τα κράτη-μέλη παίρνουν από την αρχή τη περίοδου όλο το ποσό. Το κατανέμουν στι προτεραιότητές τους, το 14-15 συγκεκριμένη φάση, και όταν ε, καθορίσαμε νέε προτεραιότητε γιατί άλλαξε η κατάσταση επιτόπου, γιατί καθορίσαμε νέε προτεραιότητες, το PNR και τέτοια, το ETIAS, ε τα κράτη-μέλη δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ανακατανομή των πόρων μεταξύ των προτεραιοτήτων, γιατί τα χρήματα είχαν ήδη δεσμευθεί. Οι αστυνομίες και οι άλλοι φορείς εφαρμογή είχαν ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή, γιατί θέλανε να προχωρήσουν γρήγορα για να έχουν αρκετό χρόνο κατά την επταετή περίοδο να ολοκληρώσουν. Αλλά όταν το 16 και το 17 καθορίσαμε νέες προτεραιότητες, είχαν ήδη δαπανηθεί ή δεσμευθεί οι πόροι Δεν μπορούσαμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την κοινή διαχείριση. Αυτό έγινε πολύ σαφώς για το ETIAS ε και για το PNR. Και άλλες ανάγκες που έπρεπε να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης και επανήλθαν στην Ένωση ζητώντας επιπλέον χρηματοδότηση. Γι' αυτό θέλουμε να υπάρχει περισσότερη ευελιξία για να ανακαθορίζουμε την κατανομή των πόρων όταν ανακαθορίζονται οι προτεραιότητες. Προχωράω καταλήγω κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, τώρα πώς λειτουργεί η διαδικασία. Κάθε δύο χρόνια θα υποβάλλετε ένα πρόγραμμα και στην Επιτροπή σας και στο Κοινοβούλιο λοιπόν και στο Συμβούλιο για τις προτεραιότητες και οι διάφορες διαδικασίες για την εφαρμογή. Θα είναι οι διεθνικές δράσεις, θα είναι η συγκροματική χρηματοδότηση προς τα κράτη-μέλη. Και αυτή η θεματική διευκόλυνση προβλέπει μία μέθοδο για να δίδονται συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις στα κράτη-μέλη, το top-up που λέμε, με πολύ ευέλικτο και μη γραφειοκρατικό τρόπο. Χρειαζόμασταν περισσότερη ευελιξία. Χρειαζόμασταν δυνατότητα να δώσουμε ένα συμπληρωματικό ποσό και να στηρίζουμε σε πραγματικό χρόνο τις πρωτοβουλίες. Γιατί αλλιώς ήταν μακροσκελής η διαδικασία αναθεώρησης των εθνικών προγραμμάτων. Ήταν πολύ περίπλοκο το σύστημα για την ε, απόδοση για την ε, εξασφάλιση συμπληρωματικής χρηματοδότησης και κατόπιν της κατανομής της στα εθνικά προγράμματα. Γι' αυτό κάνουμε κάποιες προσαρμογές για να πηγαίνουμε πιο γρήγορα. Μία άλλη βελτίωση. Υπήρξε εναρμόνιση των κανόνων με τα διαρθρωτικά ταμεία υποβάλαμε και σε εσά και σε όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους ένα εγχειρίδιο κανόνων για τα ταμεία μικτής διαχείρισης. Ούτω ώστε και οι δικαιούχοι και τα κρατημέλη να έχουν ένα σύνολο κανόνων και για το δικό μας ταμείο και για τα διαθροτικά. Για παράδειγμα, όταν θέλουμε να προστατεύσουμε δημόσιους χώρους. Άρα κάποιος, για παράδειγμα, μπορεί να έχει ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ε, ριζοσπαστικοποίησης μια συγκεκριμένη κοινότητα. Μπορεί να λάβουν χρηματοδότηση και από το δικό μας ταμείο και από τα διαθροτικά με βάση τους ίδιους κανόνες. Γιατί υπήρξαν επικρίσεις. Βέβαια ότι και πάλι αλλάζετε τους κανόνες. Ναι, τους αλλάζουμε. Αλλά τους αλλάζουμε γιατί θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη εναρμόνιση στις περαιτέρω εργασίες μας, εργασίες μας και περισσότερη απλούστευση. Εδώ βλέπετε πόσα μέσα μπορούν να συμβάλλουν στην ασφάλεια. Λοιπόν, είναι η τελευταία διαφάνεια, πρόεδρε. Τελευταία, τελευταία. Σε δύο τομείς κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Διάφορες υπηρεσίες της Κομισιόν για να εντοπίσουμε μάλλον συγγνώμη, για να καθορίσουμε ότι η ασφάλεια είναι απόλυτη προτεραιότητα και βεβαίως επειδή έχουμε και τα μέσα που χρηματοδοτούν δράσεις σε πολλές ε, τρίτες χώρες αλλά και τα δικά μας μέσα θα μπορούν να χρηματοδοτούν δράσεις σε τρίτες χώρες αλλά κυρίως ε, η χρηματοδότηση αυτών των ενεργειών θα γίνεται από τα εξωτερικά ταμεία. Έχουμε συνεργασίες και με τα προγράμματα της, ε, του Κοινωνικού Ταμείου, με το Horizon Sin και σας ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε που σας πιέζω με το χρόνο, αλλά έχουμε πάρα πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη με το απόγευμα. Ρομπέρτα, ευχαριστώ πολύ, Κλοντς. Εγώ Είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τη Μόνικα Χολμάιερ που ως εισηγήτρια δεν μπορούσε να παραβρεθεί σήμερα η οποία επιθυμεί να ευχαριστήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια πολύ ισορροπημένη πρόταση η οποία καλύπτει όλα τα θέματα και να την ευχαριστήσει και για την πολύ διεξοδική παρουσίαση που έκανε σήμερα. Εμείς καταλαβαίνουμε το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως προτεραιότητα τα θέματα ασφάλειας και προτείνει να διπλασιάσει στα 2,5 δις ευρώ τα κονδύλια για τα θέματα ε, της ασφάλειας. Και αυτό το ζητά εδώ και καιρό το ΕΛΚ. Και το γεγονός πως θέλει να ενισχύσει τα συστήματα πληροφορικής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να υπάρχει διαλειτουργικότητα και να έχουμε περισσότερες δυνατότητες ε, κατάρτισης είναι ε, κάτι το οποίο βρίσκουν σύμφωνοι την εισηγήτρια. Επίσης, Καλό είναι που συνεργαζόμαστε περισσότερο με τα υπόλοιπα ταμεία, τα ταμεία για τα σύνορα, τα ταμεία για το άσυλο και όλα τα υπόλοιπα μας παρουσίασαν, περισσότερο συνέργειες και πολλές δυνατότητες βελτίωσης εάν συγκριθούν με τις σημερινές δυνατότητες που δίνει νομοθεσία. Πλούστευση διαδικασιών και ελαχιστοποίηση του διοικητικού κόστους. Επίσης, οι διατάξεις και οι κανονισμοί που έχουν κοινέ χρηματοδοτικές διατάξεις για τα βασικά ταμεία θα αποτελέσουν κομβικά σημεία και ελπίζουμε πως οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Ρέτζι θα δημιουργήσουν ένα εργαλείο ισχυρό για να καλύψει τα θέματα αυτά. Επίσης, το γεγονός που θα διαχειρίζονται από κοινού τα κονδύλια αυτά και τα ταμεία αυτά τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ναι, και 60% στα εθνικά, στους εθνικούς προϋπολογισμούς, ναι, πολύ σημαντικό. Θα πρέπει η χρηματοδότηση αυτή να δίνεται στα κράτη-μέλη στην αρχή της προγραμματικής περίοδου και να επαναξιολογούνται στα πλαίσια τη ενδιάμεση αναθεώρησης έτσι ώστε να έχουμε ως καλύτερα αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε και έναν μηχανισμό που θα προκρίνει αυτού οι οποίοι είναι αποτελεσματικοί έτσι ώστε η προτεραιότητά μα θα είναι να επιτυχάνουμε του στόχου των προγραμμάτων και να μην παρακολύουμε με υπερβολική γραφειοκρατία. Έχουμε μια σειρά από ερωτήσει που θέλουμε να απευθύνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορώ να τα διαβάσω τώρα αν δεν σα πειράζει και θα πρέπει να συζητήσουμε επίση πω ο κανονισμός αυτός θα εξασφαλίζει πως η χρηματοδότηση θα στραφεί προς προτεραιότητες εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την απαραίτητη όμως ευελιξία που είναι σημαντικό για τα μικρά κράτη που έχουν συγκεκριμένα προβλήματα όπως εμείς την ε, Μάλτα και το νησί ε, Γκότζο για παράδειγμα. Τώρα, ποια είναι η λογική που κρύβεται πίσω από την αρχιτεκτονική των προγραμμάτων ε, στον χώρο της εσωτερικής ασφάλειας και δικαιοσύνης. Και γιατί το κομμάτι που είναι σε αποθεματικό είναι στα πλαίσια των κοινων των διατάξεων παρόλο που ε, συμπεριλαμβάνει προτάσεις και από άλλα ταμεία. Και γιατί δεν έχουμε ε, κάπου την επίγουσα ανάγκη. Πώς θα χρηματοδοτηθεί στην πράξη αυτή λοιπόν. Δώστε μας κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα για την απλούστευση διαχείριση των ταμείων και δεδομένου ότι έχουν μεγάλο ρόλο στο να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των Ευρωπαϊκών Πολιτών γιατί έχετε αποκλείσει ρητά τις, υπηρεσί, τις υπηρεσίες στον χώρο ΔΕΗ από τα ταμεία αυτά εκτός από τις περιπτώσεις επίγουσας ανάγκης. Και τέλος, τι συμβαίνει στις περιπτώσεις όπου έχουν απορροφήσει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη πριν την ενδιάμεση αναθεώρηση. Ευχαριστούμε λοιπόν και μια φορά ακόμα για το πολύτιμο αυτό σχέδιο που καταθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συνεργαστεί η Μόνικα με όλους τους σκιώδεις και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο χώρο αυτό. Ωραία, θα δώσω τώρα την Κυριακή, στην Κυριακή Έγγελ το λόγο που είναι οι σκιώδης από τους σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ, Κλόντο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή που μας παρουσίασε με ε, ξενοχιστικό τρόπο την πρότασή της και ευχαριστώ την εισηγήτρια που μας έχει ήδη προμηθεύσει με ένα πλαίσιο ε, σε σχέση με τις ε, τροπολογίες της. Είμαι βεβαία ότι θα έχουμε την μέγιστη συνεργασία όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας που είναι διαρκώς υπό εξέλιξη και που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Ακούσαμε διάφορες προτάσεις που και κριτήρια που θα υιοθετηθούν για την εφαρμογή αυτού του ταμείου όπως η η απλοποίηση, η ευελιξία και η συντονισμένη προσέγγιση. Υψηλό επίπεδο ε, συνεργασίας ε, το εγγυόμαστε όχι, ε, μάλλον και το εγγυόμαστε όχι μόνο με μέτρα αντιμετώπισης αλλά και με μέτρα πρόληψης και με συντονισμό. Γι' αυτό και τα, για τα κρατη αυτή η πολιτική είναι πολύ σημαντική για να αντιμετωπίσουμε αυτές τι κοινέ προκλήσεις. Σε ναι. αυτό προστίθεται και η ενισχυμένη ε, συνεργασία με τις τρίτες χώρες και ε, κυρίως για να ενισχύσουμε την αντιμετώπιση του θέματο ε, τη εμπορίας ανθρώπων και, μετα... και των μεταναστών και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ρεζοσπαστικοποίησης. Για μας είναι πολύ σημαντικό, ωστόσο, μέσα σε όλα αυτά να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανθρώπινη εξωπρέπεια. Το Ταμείο αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί και να εφαρμόζεται με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα που θεσπίζονται από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ένωση και ε, τι διεθνεί μα υποχρεώσει. Επίση, όσον αφορά την πτυχή τη σεβασμού των ε, δικαιωμάτων, θα εστιάσουμε την προσοχή μα. Ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια και είμαι βεβαία ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία στο εγγύηση μέλλον. Για την ώρα, λέει, δεν δεν έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ε, ε, αποσαφηνίσουμε πολλά στοιχεία που ήδη υπογραμμίστηκαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σεσίλ. Άλλος. Ωραία. Ο κύριος Γκαστέλου, λοιπόν, θέλετε να απαντήσετε σε ερωτήσεις που ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ και στην ευκαιρία που μου δίνετε να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις για τα πρώτα που ακούσαμε. Μας ρωτήσετε τι θα γίνει αν τα κράτη-μέλη έχουν απορροφήσει όλα τα κονδύλια πριν την ενδιάμεση αναθεώρηση. Ακριβώς γι' αυτό έχουμε τις θεματικές διευκολύνσεις, τους μηχανισμούς αυτούς, έτσι ώστε κάθε δύο χρόνια, δηλαδή το 2021, το 2023, το 2025 και το 2026, που ίσως είναι λίγο αργά, για την αναδιανομή. έτσι ώστε και μετά την ενδιάμεση αναθεώρηση να στηρίξουμε και τις νέες προτεραιότητες. Παραδείγματα απλούστευσης. Κάτι που δεν χρησιμοποιήσαμε για παράδειγμα στο παρελθόν ήταν η, η απλουστευμένη καταποκοπήν χρωματοδότηση, κάτι το οποίο δίνει μεγάλη ευελιξία στα κράτη-μέλη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα, όχι γιατί δεν είναι ελκυστικό, αλλά γιατί τα κράτη-μέλη φανταζόντουσαν πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στείλει πιο ξεκάθαρη πιο ξεκάθαρες οδηγίες στο θέμα αυτό. Αυτό που θα κάνουμε είναι να μην χρειάζεται να ορίζονται αρμόδιες αρχές έτσι ώστε να ξεκινήσουν να εφαρμόζουν από την πρώτη μέρα τα κρατημέλη αυτά τα κονδύλια χωρίς να χρειάζεται να ορίσουν την αρχή ε, ελέγχου ή διαχείρισης. Θα γίνονται οι εκ των υστέρων έλεγχοι βεβαίως, έτσι ώστε οι αρχές που ε, κάνουν τη δουλειά σου να τον κάνουν σωστά, αλλά θα γίνεται πιο γρήγορα. Τώρα, για το τι δεν επιτρέπεται οι υπηρεσίες ε, στην επίγουσα έκτακτη βοήθεια ε, να χρηματοδοτούνται. Γιατί θέλουμε να έχουμε έναν οργανωμένο προπολογισμό, είστε εσεί η δημοσιονομική μα αρχή και θέλουμε να έχουμε ξεχωριστέ γραμμέ χρηματοδότηση, άλλε για τα εργαλεία μα και άλλε για τι υπηρεσίε. Γιατί αν ξεκινήσουμε να επιτρέπουν τη μεταφορά κονδυλίων από το Ταμείο ε, για την Ασφάλεια προ τι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τι εξωτερικέ υπηρεσίε, τότε δεν θα είναι εύκολο για εσά να τα παρακολουθήσετε. Γιατί εσεί έχετε και το ρόλο αυτό τη παρακολούθηση και νομίζω πως από την αρχή είχαμε πει ότι αυτά θα μοιραστούν και θα λέμε τόσα για τα ταμεία ασφάλειας, τόσα για τις υπηρεσίες. Τώρα, για το κατά πόσο αν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από Αυτέ τι αρχέ για την έκτακτη βοήθεια, ναι, μπορούμε να το κάνουμε, γιατί έχουμε συμφανίσει ότι για τι επίγουσε ανάγκες μπορεί να χρειάζεται ταχύ ανάληψη δράση, οπότε εκεί μπορούμε να παρεκκλίνουμε από τη βασική ιδέα που είχε η αρχή, η δημοσιονομική, η οποία εξασφαλίζει την αρχή τη παρακολούθηση. Τώρα, το πώ θα λειτουργήσει η έκτακτη βοήθεια, πολύ σπάνια έχει χρησιμοποιηθεί για την ασφάλεια, έχει χρησιμοποιηθεί για, ε, για το προσφυγικό, για τα σύνορα, αλλά όχι για την ασφάλεια. Θα πρέπει αυτά να περιορίζονται στο ελάχιστο γιατί θεωρούμε πως θα πρέπει να είναι οι θεματικοί μηχανισμοί για να προσθέσουν στη χρηματοδότηση όπου χρειάζεται αλλά αυτή η επίγουσα βοήθεια θα εστιάζεται όπως και τώρα σε αίτημα από το κράτος μέλος και κάθε φορά θα αποφασίζει κατά περίπτωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θα χορηγήσει ή όχι, βασιζόμενοι και σε πρόγραμμα εργασία και βεβαίω κοινοποιώντα όλα αυτά ε, μία φορά κατ' στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μέχρι σήμερα την επίγουσα ανάγκη την έδινε απευθεία ε, σε ενδιαφερόμενο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να είναι η Europol, κάποιο ε, άλλο όργανο. Τώρα θα πηγαίνει στο κράτος μέλος έτσι ώστε να εφαρμόζει τη χρηματοδότηση αυτή το κράτος μέλος. Ενώ μέχρι τώρα στο παρελθόν η εφαρμογή γινόταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε διοικητικά, διαχειριστικά την έκτακτη βοήθεια θα μπορεί να την αναλαμβάνει το κράτος μέλος εφόσον έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτήματος και κατάθεσης προγράμματος εργασίας. Για το 10% και το αποθεματικό να σας πω πως τα διαστροτικά ταμεία δεν έχουν ε, τέτοιου είδους ε, πλαφόν. Η εμπειρία μας με το 10% στο παρελθόν δεν ήταν πολύ καλή, αλλά θεωρούμε πως εδώ, αντίθετα με το τι συμβαίνει στα διαστροτικά ταμεία, χρειαζόμαστε να είμαστε πολύ περισσότερο ευέλικτοι. Ο δικός μας χώρος χρειάζεται ευελιξία, χρειάζεται ε, να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε μια μεταλλασσόμενη πραγματικότητα, οπότε θα πρέπει να μπορούμε να προσαρμόσουμε και γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται μια αναδιανομή ε, στην αναθεώρηση και γι' αυτό έχουμε αυτό το 10% όπως σας είπα μέσα στο αποθεματικό. Στα διαφορετικά ταμεία ε, τα πράγματα είναι διαφορετικά, η κατάσταση επιτόπου δεν είναι τόσο ρευστή, οπότε δεν χρειάζονται αυτού του είδους την ευελιξία. Και για τις τρίτες χώρες που ακούσαμε μια ερώτηση, όντως, εδώ έχουμε μια αλλαγή και στο Ταμείο Ασφάλειας, όπου έχει στηθεί το Ταμείο έτσι ώστε οποιαδήποτε δράση μπορεί να γίνει εσωτερικά, να μπορεί να γίνει και εξωτερικά σε τρίτη χώρα. Γίνεται υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει. Θεωρούμε πω αυτά τα εξωτερικά εργαλεία είναι τα καλύτερα στα οποία θα πρέπει να επενδύσουμε για να αναλαμβάνουν δράση για τέτοιου είδου έργα σε τρίτε χώρε. Και αν δεν δρούν τα εξωτερικά εργαλεία θα μπορούσαμε εμεί μέσω του Ταμείου ε, εσωτερική ασφάλεια, να αναλαμβάνουμε και εμεί δράση χάρη σε αυτές τις νέε διατάξει. Τώρα, για τι θεμελιώδει ελευθερίε και τα ανθρώπινα δικαιώματα Έχουμε δύο διατάξεις στον κανονισμό για την προστασία αυτών, με την επιφύλαξη βέβαια του συστήματος αξιολόγησης και αναφοράς. Γιατί αυτά τα προσέχουμε ιδιαίτερα το ίδιο κάνουν και τα κράτη-μέλη και μέχρι σήμερα νομίζω ότι ήταν πολύ ε, επιτυχημένη η παρακολούθηση των θεμάτων αυτών στα πλαίσια τη ασφάλεια αλλά και των συνόρων και τη μετανάστευση. Είμαστε λοιπόν πολύ ευχαριστημένοι από το πώ έχουν δράσει οι διατάξει για τι θεμελιώδει ελευθερίε και τα ανθρώπινα δικαιώματα και βέβαια πώ συνδυάζονται και με τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτά αν έχετε και άλλες ερωτήσεις να απαντήσω και σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας τα παρουσιάσω. Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Πρέπει να κλείσουμε με το σημείο αυτό. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Θα περάσουμε τώρα στο σημείο 6 που είναι το σύστημα ε, εισόδου-εξόδου με τις δύο διορθώσεις στο κείμενο. Ο κύριος Δίας Δεμέρα δεν είναι εδώ σήμερα Οπότε θα σας πω ποια είναι τα τρία μικροζητήματα τα οποία καλύπτει αυτό το διορθωτικό. Να τα διαβάσω για να καταγραφούν. Πρώτη διόρθωση. Για όσους έχουν ε, διαβατήρια Αγίας Έδρας, που δεν καλύπτονται από το Βατικανό, ε, που δεν ε, καλύπτονται από τον κανονισμό, πρέπει λοιπόν να ε, τους προσθέσουμε είναι οι πολίτες Βατικανού. Επίσης το 32 αναφέρεται σε τους μόνιμα διαμέναντους και σε αυτούς ε, θα πρέπει να διαγράψουμε το if applicable και τις αγγίλες στο τέλος της πρότασης. Και από εκεί να πάει η αγγείλη στην αρχή της πρότασης, έτσι ώστε να φαίνεται ότι καλύπτει όλα τα σημεία. Είναι τεχνικά τα ζητήματα αυτά, αλλά θα πρέπει να το διορθώσουμε. Τα έχετε και μπροστά σας. Ο κύριος Δίας Δεμέρα θεωρεί πως δεν υπάρχει πρόβλημα και θα πρέπει η Επιτροπή μα να τα δεχτεί. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλετε κάτι να πείτε? Εάν όχι... Καταλήγω λοιπόν πως εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θεωρούμε ότι σύμφωνα με τον κανόνα 2.3.1 γίνονται δεκτά αυτά τα διορθωτικά σημεία ε, και καταγράφεται αυτό και σύμφωνα και με τον κανόνα 2.31 παρένθεση 4 θα το ανακοινώσουμε και στην Ολομέλεια. Περνάμε στο σημείο 7. Έχουμε το σχέδιο γνωμοδότησης για την έκθεση Γιούρι για την προστασία των ανθρώπων που καταγγέλουν παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας. Μάιτε, η Μάιτε είναι η συγγήτρια, δεν είναι όμως εδώ σήμερα. Ο κύριος Ντεπρέ θα παρουσιάσει στη θέση της τη γνωμοδότηση αυτή. Ζεράρτ. σε ευχαριστώ που το έκανες. Έχει το λόγο εκ μέρους του Μάιτε. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ζητά συγγνώμη, συνάδελφός μου, Μάιτε Παγαθαουρτούντουα, που δεν μπορεί να παρευρεθεί, γιατί έχει υποχρεώσεις εκτός Βρυξελών εκ μέρους της θα σας παρουσιάσω τη γνωμοδότηση που προτείνει για την πρόταση οδηγίας για την προστασία των ατόμων που καταγγέλουν παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου. Επίσης τονίζει Μάιτε ότι συνεργάστηκε στενά με την κυρία Ροζιέρη την εισηγήτρια της Επιτροπής ε, Τζούρι και συμφώνησαν το σχέδιο γνωμοδότησης να συμπληρώσει το σχέδιο έκθεσης που θα υποβληθεί στη Τζούρι. Οι τροπολογίες που αφορούν τη διαδικασία καταγγελιών είναι ελάχιστες. Οι δύο εισηγήτρες θεωρούν ότι η Κομισιόν ή ότι Επιτροπή Τζούρι πρέπει να ασχοληθεί η εισηγήτριά μας προτείνει ορισμένες τροπολογίες που συμπληρώνουν και κάνουν πιο συνεπή την πρόταση, ιδιαίτερα προσθέτοντας ε, κριτήρια ερμηνείας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τον ορισμό του εργαζόμενος. Δεύτερον, μια άλλη ιδέα επί της οποίας επιμένει ιδιαίτερα η εισηγήτριά σας είναι ότι πρέπει να αυξηθεί η προστασία των καταγγελόντων και εκτός του περιβάλλοντος εργασίας. Οι πιο άμεσες και οι πιο αρνητικές επιπτώσεις γενικά βέβαια προκύπτουν όταν υπάρχει ε, σχέση εργασίας. Αλλά η συγκίτρια τονίζει ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο ιδιωτικό βίος του καταγγέλλοντος μπορεί να θυγεί σοβαρά από αυτά που συμβαίνουν στον χώρο εργασίας. Πρέπει λοιπόν η προστασία να επεκταθεί και προς αυτή την κατεύθυνση και προτείνονται διάφορες τροπολογίες ούτω ώστε να συμπληρωθεί η προστασία των ατόμων αυτών. Τρίτον, μια άλλη ιδέα που προτείνεται στις τροπολογίες είναι ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανωνύμων καταγγελιών, όχι απλώς εμπιστευτικότητα. Εάν το σύστημα της εμπιστευτικότητας δεν αρκεί για την προστασία, η ανωνυμία ίσως να είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσει ένα άτομο την προστασία του. Η εισηγήτριά μας περιλαμβάνει και ορισμένους ορισμούς από τον νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων για να υπάρξει περισσότερη νομική ασφάλεια και για να διευκολυνθεί η διαμεθοριακή ασφάλεια των καταγγελόντων και πρέπει να περιορίζεται η συλλογή στοιχείων που δεν έχουν καμία σχέση με τους στόχους της οδηγίας. Καταλήγοντας, το σχέδιο γνωμοδότησης της ε, εισηγήτριάς μας περιέχει 32 τροπολογίες που όπως είπα προσπαθούν να επιτύχουν μια ισορροπία με όσα θα προτείνει η κυρία Γοζιέρ στην Τζούρι. Η εισηγήτριά μας καταλήγοντας τονίζει ότι έχει κάθε βούληση και διαθεσιμότητα για συνεργαστεί με όλους τους σκιώδεις για να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Ζεγά. Θαυμάσια παρουσίαση. Με τόση θέρμη θα μπορούσε να ήταν δική σας η γνωμοδότηση. Λοιπόν, η κυρία Στίβενς θέλει να μιλήσει από πλευράς του ECR. Ε, ε Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εργασία της. Η πρόταση αυτή κυρίως αφορά την τζούρι, αλλά χαίρομαι που μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε. Υπήρξαν πρόσφατα σκάνδαλα, το Dieselgate, το, οι διαρροές του Lux, το Leaks, το Cambridge Analytica, τα έγγραφα του Παναμά, αυτό καταδεικνύει ότι οι καταγγέλλοντες παίζουν ζωτικό ρόλο για να αποκαλύπτονται παράνομες πρακτικές που θίγουν και τους πολίτες και την κοινωνία μας. Οι καταγγέλλοντες είναι εγγυητές της διαφάνειας. Πρέπει λοιπόν να τους προστατεύσουμε. Όμως ε, η οδηγία έχει ένα πολύ ευρύ ορισμό για τον όρο καταγγέλλοντες, whistleblower. Και αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ότι δεν παρέχεται επαρκής ε, προστασία στους πραγματικούς καταγγέλλοντες. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα συμφέροντα των εργοδοτών. Πρέπει λοιπόν να παρέχουν οι καταγγέλλοντες αποδείξεις αυτών τα οποία ισχυρίζονται. Μπορούμε να συνεργαστούμε για να υπάρξει ένα καλό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κώστα από πλευρά των σοσιαλιστών. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε για την γνωμοδότηση και την εργασία μέχρι τούδε της ε, εισηγήτριας. Χάρη στην επιμονή του Κοινοβουλίου τελικά η Επιτροπή πρότεινε ένα νομοθετικό κείμενο. Όλοι συμφωνούμε ότι επιτέλους είναι ώρα για να προστατευθούν οι καταγγέλλοντες παραβιάς του ε, ενωσιακού ε, δικαίου. Για τους σοσιαλιστές είναι σαφές ότι οι καταγγέλλοντες παίζουν ζωτικό ρόλο για να αποκαλυφθούν παράνομες πρακτικές και συμπεριφορές. Είναι ουσιώδης ο ρόλος τους για την προστασία του κοινού συμφέροντος, για να διασφαλίζεται η διαφάνεια, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της φοροδιαφυγής, είναι ουσιώδης πυλώνας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ούτως ώστε οι πανίσχυρες επιχειρήσεις και κυβερνήσεις λογοδοτούν. Έτσι πολλές μυστικές προφορίες ε, βγαίνουν στο φως. Αλλιώς αυτές οι πληροφορίες θα έμεναν στο σκοτάδι. Είναι αναγκαία λοιπόν η λειτουργία τους για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την ελεύθερη διαμόρφωση γνώμης. Καλωσορίζω την πρόταση της εισηγήτριας που ενισχύει την ανωνυμία και εμπιστευτικότητα και έτσι βελτιώνει την πρόταση της Επιτροπής. Τέλος, τονίζω ότι οι καταγγέλλοντες δρούν υποκείμενοι σε πολύ υψηλούς ατομικούς και οικονομικούς κινδύνους και πολύ συχνά πληρώνουν βαρύ τίμημα. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς μπορούμε να τους αποζημιώσουμε. Τι μορφή θα μπορούσε να έχει κάποια ανταπόδοση. Προσβλέπω στην καλή συνεργασία με την εισηγήτρια. Έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι και είμαι πεπισμένος ότι θα καταλήξουμε σε ικανοποιητικές λύσεις για ισχυρή προστασία των ατόμων που καταγγέλουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου. Ευχαριστώ, Ντίτμαρ, λέει ο Πρόεδρος. Μπάρμπαρα Σπινέλη. Ε, Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική τη εργασία και για τι τροπολογίε τη για την προστασία των δεδομένων και τι ανωνυμίε, ώστε να εγγυηθούμε στου μάρτυρε δημοσίου συμφέροντο που το επιθυμούν να μην αποκαλύπτουν την ταυτότητά του. Οι τροπολογίε μου θα αφορούν κάποιε επιπλέον πτυχέ που θα μπορούσαν ίσω να βελτιώσουν την πρόταση που ήδη είναι πολύ αξιέπαινη ω βάση κίνηση. Γι' αυτό το σκοπό θα υποβάλω τροπολογίε που στόχο θα έχουν να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας και να μην περιορίζεται στις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της πρότασης. Κατά συνέπεια, ο κατάλογος των διατάξεων μπορεί να, να, είναι πιο ευέλικτος ή και να καταργηθεί. Και να προσθέσουμε εκεί την φράση ευρωπαϊκή ε, διατάξεις ή νομοθεσίες. Επίση, θεωρώ πω αυτή η οδηγία θα πρέπει να προσφέρει την προστασία τη στου ανθρώπου που διευκολύνουν την ε, παρουσίαση αυτών των πληροφοριών, δηλαδή διάφοροι διαμεσολαβητέ ή ε, δημοσιογράφοι έρευνα που με τι δραστηριότητέ του μπορούν να εγγυηθούν την διάδοση αυτών των πληροφοριών ή την αποκάλυψη αυτών. Προστασία θα πρέπει να έχουν δε και οι φοιτητέ, ερευνητέ, οι εργαζόμενοι, οι πρώην υπάλληλοι, καθώς και οι διάφοροι σύνδεσμοι. Σημαντικό σημείο επίση προτεραιότητα είναι η δυνατότητα του ε, μάρτυρα δημοσίου συμφέροντο να επιλέγει τον διάβλο που, ε, που θα χρησιμοποιήσει για να κοινοποιήσει τα στοιχεία που έχει, να καταργηθεί το ιεραρχικό σύστημα, δηλαδή πρώτα εσωτερικά ε, εσωτερική ιεραρχία και μετά εξωτερική που προτείνει η Κομισιόν. Και ε, έχω το εξή ερώτημα ουσία. Μήπω δηλαδή θα έπρεπε να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή αυτή τη οδηγία και στου ευρωπαϊκού θεσμού και στο σύνολο των οργανισμών τη Ένωση, όχι μόνο αυτού που απαριθμούνται στην πρόταση, στο βαθμό που μπορεί να ε, έχουν να κάνουν με δραστηριότητε ε, μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στην εφαρμογή τη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα ήταν πολύ σημαντικό μήνυμα στους ε, πολίτες που αυτή τη στιγμή δυσπιστούν απέναντι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε μεγάλο βαθμό. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την σας, τις εμπεριστατωμένες σας απαντήσεις ε, και ερωτήσεις. Ε, θα τις διαβιβάσουμε στην εισηγήτρια. Ήθελες εσύ, Ζεράρ, να προβείς σε συμπεράσματα. Πρόεδρε, δεν θέλω να προβαγώ σε συμπεράσματα, δεν είμαι εγώ εισηγητής, ε, ούτε σκιώδης εισηγητής. Ε, θα διαβιβάσω ε, τις παρατηρήσεις των συναδέλφων και τις ερωτήσεις και έχω την εντύπωση ότι η συζήτηση θα γίνει σε εξαιρετικό κλίμα και δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι θα έχουμε το καλύτερο δυνατό ε, αποτέλεσμα. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Και εγώ ευχαριστώ που αντικατέστησε την εισηγητή. Η προθεσμία είναι 14 Σεπτεμβρίου για την υποβολή τροπολογιών. Προβλέπεται η συζήτηση στις 10 Οκτωβρίου και την Τζούρι στις 22 ε, Οκτωβρίου. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Θα περάσουμε τώρα στο σημείο 8, κοινή συζήτηση για την διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το σημείο 8 και 9. θα εξετάσουμε τις τροπολογίες, τις δύο τροπονομοθετικές προτάσεις για τη διαλειτουργικότητα. Βλέπω πως οι εισηγητές μας είναι εδώ παρόντες. Θα δώσω το λόγο στους δύο μας εισηγητές, ο κύριος Λένας και μετά ο κύριος Μέλο. Και μετά θα ακούσουμε τους Σκιώδης. Κύριε Λένα, παρακαλώ πρώτα εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι πολύ καλό το ότι όλοι περάσαμε πολύ ωραία το καλοκαίρι μας ε, ε, στην πισίνα ή στη θάλασσα, στην παραλία, διαβάζοντας τις τροπολογίες. Λάβαμε γύρω στις χίλιες τροπολογίες για τη ε, σύνορα και τις θεωρήσεις και 926 ε, τροπολογίες για το άλλο φάκελο, δηλαδή 2.000 τροπολογία που ακούγεται πολύ, αλλά για να σας πω ε, ειλικρινά και κατά τη σύνταξη της σχεδίου έκθεσης είχαμε διαπιστώσει ότι το να κάνουμε μικρές αλλαγές αλλά να γίνουν σε ολόκληρο το, το κείμενο αυτό οδηγεί σε πολλές τροπολογίες. Δηλαδή δεν είναι η ποσότητα αλλά η ποιότητα των τροπολογιών που μετράει και είμαι βέβαιος ότι περισσότερες από αυτές θα δώσουν καλή καλή βάση δίνουν καλή βάση για τη δουλειά μας και για την περαιτέρω βελτίωση της πρότασης της Επιτροπής. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας τους κοιόδης όλων των ομάδων επειδή τροποποίησαν και τα δύο, τους δύο φακέλους με συνεπή τρόπο. Από τη φύση συνδέονται μεταξύ τους αυτοί οι δύο φάκελ και γι' αυτό και οι τροπολογίε έγιναν έτσι συντονισμένα. Ε, είμαι ευγνώμων που όλοι ε, ακολουθήσατε αυτήν την, τον τρόπο εργασίας. Η κοινή δήλωση από του τρει θεσμού ε, δείχνει αυτό το φάκελο ω πρώτης προτεραιότητα για φέτο. Ως εισηγητέ, σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε αυτή τη φιλοδοξία με φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα Έχουμε σχεδιάσει ήδη πολλές ε, τροπολογίες ε, για τις επόμενες μέρες. Τώρα σε σχέση με τις επαφές ε, και βεβαίως επειδή ε, κολούθησε τον καλοκαιρινές διακοπές στην πρώτη μας συνεδρίαση, θέλαμε να πούμε ότι θέλαμε να υπά... χρησιμοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό τα υπάρχοντα μέσα, αλλά και τις πληροφορίες που έχουμε ήδη και να μην συλλέξουμε και άλλα δεδομένα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν είναι μια ευφυής απάντηση σε αυτά τα δύο αιτήματα χωρίς να αλλάζουν τα δικαιώματα πρόσβασης, χωρίς να εγκαταλείπουμε τους κανόνες προστασίας δεδομένων, η διαλειτουργικότητα θα εξασφαλίσει ταχύτερη, πιο συστηματική πρόσβαση στα συστήματα της Ένωσης για τους επαγγελματίες, δηλαδή αστυνομικού και τους συνοριοφύλακες, ώστε να έχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται. Δεν ξέρω πόσο χρόνο μου δίνετε, Πρόεδρε, αλλά θα ήθελα να περάσω στο περιεχόμενο των τροπολογιών, διότι πιστεύω ότι εν γέννη αυτές δείχνουν ότι υπάρχει μια ευρία πλειοψηφία των ομάδων του Κοινοβουλίου ε, της βασικής αρχής της διαλειτουργικότητας ανάμεσα στα συστήματα πληροφοριών. Επιπλέον είναι σαφές ότι οι περισσότερες ομάδες προτιμούν να μείνουμε κοντά στα συστατικά αυτά ε, τα στοιχεία που προτείνει η Κομισιόν, ενώ κάνουμε και κάποιες βελτιώσεις δηλαδή καλύτερα backup, δηλαδή στήριξη, υποστήριξη, κανόνες ασφάλειας, καλύτερη παρακολούθηση, βελτίωση ε, κανόνων προστασίας δεδομένων, διόρθωση κάποιων ανακριβιών που εντοπίσαμε στη διάρκεια της συζήτησής μας ε, στην πρώτη πρόταση και ε, τροπολογίες για να βελτιωθεί και να χτιθεί το πεδίο της πρότασης. Όλα αυτά νομίζω θα μας βοηθήσουν να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες επίσης αν και αναμφίβολα κατατέθηκαν με καλές προθέσεις, φοβούμε πως θα ε, ε, υπονομεύσουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων στην πράξη. Και αυτός δεν μπορεί να είναι ο στόχος ε, της εργασίας εδώ. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως η διαλειτουργικότητα ως έννοια θα θεσπιστεί και ότι θα δουλέψουμε με τους συναδέλφους ώστε να εξασφαλίσουμε την υλοποίηση αυτού. Σας ευχαριστώ όλους. Προσβλέπουμε στην ε, συνεργασία με όλους. Δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε. Θα ξεκινήσουμε ήδη από αύριο. Να σας συγχαρώ. Για τον, να σας συγχαρώ για τον σαρκαστικό τρόπο με τον οποίο να ξεκινήσατε την εισήγησή σας, κύριε Ελένα. Πολύ αστείο μου φάνηκε, πολύ καλό. Ο κύριος Μέλο. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχα... Ελπίζω όλοι να περάσατε καλές διακοπές. Αν δεν σας πειράζει θα μιλήσω πορτογαλικά, που, πράγμα που κάνω ούτως ή άλλως σε αυτές τις συνεδριάσεις, για να σας πω λοιπόν, καταρχάς θέλω να υπογραμμίσω το μεγάλο εύρος ε, των ε, τροπολογιών που έχουν υποβληθεί ε, και δικαιολογούνται τόσο από το πολύπλοκο χαρακτήρα του θέματος όσο και από το, τους κανόνες που θέλουμε εδώ εμείς να τηρήσουμε. Έχουμε ήδη κάνει πολλές επαφές φυσικά με τους σκιώδεις, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω για την προσήλωσή τους και τη συμμετοχή τους σε αυτές τις συνεδριάσεις, καθώς και για τα θέματα τα οποία μας έθεσαν και μας οδήγησαν όλους να σκεφτούμε καλύτερα το τι διακυβεύεται. Έχουμε κάνει συνεδριάσεις ε, με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με εμπειρογνώμονες της Europol, του Frontex, του Ιούλης, ε, ε, του εκπροσώπους των διαφόρων ε, ε, αρμοδίων φορέων. Πολλές τεχνικές επίσης συνεδριάσεις έχουμε προγραμματίσει ώστε να επιτύχουμε το στόχο που επιθυμούμε. Ακριβώς θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τους διάφορους βοηθούς μας, συμβούλους, τόσο του δικού μου επιτελείου, όσο ε, και του επιτελείου του ΕΛΚ και της Επιτροπής μας εδώ γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι περίπλοκο και πολύ ιδιαίτερο. Μπορεί να αποτελέσει εφιάλτη αλλά τελικά ε, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία υπερβαίνουν τα απλά νομικά ζητήματα. Πολλέ από τι τροπολογίε που υποβλήθηκαν συμπεριλήφθηκαν στι συμβιβαστικέ προτάσει που θα συζητήσουμε. περί τίνος πρόκειται ακριβώς. Ε, εδώ. Θέλουμε να υπάρχουν γρήγορα οι απαραίτητε πληροφορίε προ τι αρμόδιε αρχέ, δηλαδή αστυνομία, ε, υπεύθυνοι των υπηρεσιών μετανάστευση έτσι ώστε οι τρομοκράτε και άλλοι εγκληματίε να μπορούν άμεσα να αντεπιστούν με βάση αυτές τις βάσεις δεδομένων. Ήδη είναι, υπάρχουν ένα σωρό βάσει δεδομένων, βά, δεδομένων οι οποίε όμω δεν είναι συνδεδεμένε μεταξύ του. Δεν είναι φυσιολογικό στοιχεία που ήδη υπάρχουν και που μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή εγκλημάτων να μην είναι διαθέσιμες ή να μην μπορεί κανείς να τις μοιραστούν οι αρμόδιες αρχές μεταξύ τους. Και ε, ακριβώς ε, στο σωστό μέτρο νομιμότητας για την κάθε ε, έρευνα που διεξάγει κάθε μια από αυτές τις μονάδες. Πρόκειται δηλαδή για ένα θέμα το οποίο λαμβάνει υπόψη την νομιμότητα και την νομιμοποίηση. Δεν είναι φυσιολογικό να διαβάσουμε τίτλους όπως αυτοί εδώ στις εφημερίδες. Δηλαδή, ένας εγκληματίας ε, τρομοκράτης είχε 14 διαφορετικές ταυτότητες. Ένας άλλος ε, κακοποιός στη Μασελία, 7 διαφορετικές ε, ταυτότητες. Στην Γερμανία ένας άλλος τρομοκράτης ήταν γνωστός με τέσσερις διαφορετικές ταυτότητες. Δεν είναι φυσιολογικό να επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τρομοκράτες που μπαίνουν, να μπαίνουν να επιτίθενται εναντίον μας και να ε, σκοτώνουν Ευρωπαίους πολίτες. Και αυτό οφείλουμε να το καταπολεμήσουμε. Τέλος, θέλω να σας πω ότι πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο θέλουμε ως πολιτική. Είτε θα πρέπει να διευκολύνουμε τη ζωή των ε, τρομοκρατών, είτε να την, να την ε, δυσκολέψουμε. Ως πολιτική, λοιπόν, πρέπει να νομοθετήσουμε προς την κατεύθυνση της, ε, του να κάνουμε τη ζωή δύσκολη στους τρομοκράτες και στους εγκληματίες. Γιατί, στην Ευρώπη, γιατί θέλουμε μια Ευρώπη που προστατεύει και που υπερασπίζει την ιστορική της ασφάλεια, με σεβασμό βεβαίως στα ατομικά δικαιώματα και τη την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η προστασία της ζωής και της εσωτερικής μας ασφάλειας είναι προτεραιότητα και με αυτό το στόχο ως εισηγητής δουλεύω σε αυτή την έκθεση. Πιστεύω ότι στο τέλος θα έχουμε ένα αποτέλεσμα καλό που θα λαμβάνει υπόψη τι διάφορες ευαισθησίες των διαφόρων ομάδων. Είμαι βέβαιος πως όλοι μας έχουμε τον ίδιο στόχο. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια των πολιτών με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα. Πολύ φιλόδοξο το ε, χρονοδιάγραμμα, αλλά θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μέλο και ευχαριστώ που αναφέρατε το, τους συνεργάτες μας Σα ευχαριστώ και του δύο και βεβαίω εύχομαι καλή επιτυχία γιατί έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας. Εφόσον είναι τόσο πολλέ τροπολογίε. Αλλά δεν μιλήσατε πολύ για το περιεχόμενο των τροπολογιών. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια αρχική συζήτηση για τα θέματα αυτά, γιατί έχουμε πολλού κοιόδε. Κύριε Νίντο Μίλλερ, θέλετε να κάνετε κάποιε αρχικέ παρατηρήσει για, το, ε, ε, για του σοσιαλιστέ να εκπροσωπώ την Μίρια Μντάλη επίσης, που είναι ισκιώδης για τη διαλειτουργικότητα, για την αστυνομική και δικαστική αστυνομική για τα θέματα ασύλου και μετανάστευσης. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ τους συναδέλφου. Σίγουρα ήταν πολύ σκληρό το καλοκαίρι σας γιατί δουλέψατε για την διαλειτουργικότητα. Σας ευχαριστώ για αυτό. Κάποιες αρχικές σκέψεις για τις τροπολογίες. και κατόπιν θα αναφερθώ και στις δικές μας τροπολογίες. Από την αρχή έχουμε μερικές ε, μεγάλων ε, διαστάσεων ανησυχίες γιατί θεωρούμε ότι ε, διακυβεύονται μερικά βασικά δικαιώματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων, γιατί υπάρχει κίνδυνος όλο και πιο εύκολης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, είτε από αυτά τα συστήματα ή από τα νέα ε, συστατικά διαλειτουργικότητας. Η απο τα νεα συστατικα χρήσης και αποθήκευσης αυξάνεται και η δυνατότητα να επιδιώξει κανείς δικαστική ε, ε επίλυση είναι περιορισμένη. Δεν υπάρχουν ε, επαρκείς ε, διαφυλάξεις. Η διελτουργικότητα αυτών των ε, τραπεζών δεδομένων, φάσεων δεδομένων, μπορεί να δώσει κάποια ωφέλη, αλλά έχει και πολλά αρνητικά και ξέρετε όλοι ότι από την αρχή η ομάδα μας είχε πολλές ανησυχίες, αλλά δεν είναι μόνο δικές μας ανησυχίες. Τη συμμερίζεται και η αρχή θεμελιδών δεδομένων, ο Επιτρεπτής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 και πολλέ άλλες επιτροπές και πολλά άλλα κόμματα στο σώμα. Για να μειωθούν οι κίνδυνοι που περιέχονται στην πρόταση τη Κομισιόν, υποβάλλαμε μια σειρά τροπολογίες σε στενή συνεργασία ε, με τη Μύριαμ, εγώ και η Μύριαμ, δηλαδή συνεργαστήκαμε. Γενικά θέλουμε να είμαστε αυστηροί με την διαλειτουργικότητα όπως μας την παρουσίασε ο Επίτροπος. Δηλαδή η δυνατότητα συνεργασίας και ανταλλαγής προφοριών μεταξύ βάσεων δεδομένων. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να μην είναι τόσο διευρυμένη για να συμπεριλάβει και κάποιους άλλους συμπληρωματικούς στόχους που δεν είναι αναγκαίοι και αναλογικοί και να συνδεθούν και άλλες βάσεις δεδομένων. Υπάρχουν τρία δομικά θέματα που θεωρούμε ότι είναι βασικά ως ομάδα. Είναι η απάλληψη των βιομετρικών στοιχείων, η απάλληψη του κοινού, της κοινής ταυτότητας και πρέπει να εμείνουμε στους βασικούς κανόνες για τα υποκείμενα συστήματα, για το κοινό ε, για την κοινή βάση προσωπικών δεδομένων θεωρούμε ότι δεν προσφέρει, δεν προσφέρει τίποτα καινούργιο, δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί. Για να εντοπίσουμε και να ταυτοποιήσουμε σωστά υπηκόους τρίτων χωρών αρκεί να έχουμε τα στοιχεία στις υποκείμενες ε, βάσεις δεδομένων και με βάση την χρήση των βιομετρικών και συνδέοντας χωριστά τις διάφορες υποκείμενες βάσεις με τον ε, ανοιχτευτή ταυτότητας. Δεν χρειάζεται τα ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία όλων των ατόμων να τα έχουμε και σε ένα σύστημα και σε όλες τις υποκείμενες βάσεις. Αυτό δεν σέβεται τις αρχές του κανονισμού προσωπικών στοιχείων. Και δεν είμαστε η μόνη πολιτική ομάδα που το πιστεύει αυτό. Επίσης, στις τροπολογίες μας λέμε ότι η υπηρεσία για την κοινή βιομετρική ε, αναζήτηση θα πρέπει να μην αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών, των προσωπικών δεδομένων γιατί αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν να, για να καθοριστεί ένα άτομο. Γιατί ε, σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε τις ανησυχίες που ε, ανέφερα και προηγουμένως. Επίσης, η πρόταση Η πρόταση ε, δεν διασφαλίζει ότι οι αναζητήσεις που θα γίνονται παρέχουν εγγυήσεις ότι είναι αναγκαίες και περιέχουν σοβαρές παραβιάσεις της αρχής της ε, στοχευμένης αναζήτησης. Και έχουμε και άλλες τροπολογίες για την πολιτική ταυτοποίηση, τους διάφορους ε, συνδέσμους που υπάρχουν στον ανοιχτευτή ταυτότητας. Θέλουμε να βελτιώσουμε επίσης τη δυνατότητα να προσπαθεί κανείς να διορθώσει τα στοιχεία του. Είμαστε πεισμένοι ότι οι εισηγητές θα κατανοήσουν τις ανησυχίες μας και ότι θα λάβουν υπόψη τις βασικές προτάσεις μας, ούτως ώστε να έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα που είναι αποδεκτό από όλους και προσβλέπουμε σε μια επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα την κυρία Νταλή και στον άλλο φάκελο. Επειδή έχουμε ψηφοφορίες στις 6, θα ήθελα μόνο οι σκιώδες να πάρουν το λόγο. Η κυρία Έρνστ εκ της Ζεράρ, είστε σκιώδης. Ναι, οπότε θα πάρετε το λόγο. Κορνίλια, εκτός μικροφώνου. Ποιος λοιπόν θα μιλήσει πρώτος. Ζεράρ και μετά η Κορνίλια. Δεν ζήτησα να μιλήσω πρώτος. Απλώς ήθελα να σε πιστήσω την προσοχή στο ότι είμαι σκιώδης, ο μόνος από την ομάδα μου, οπότε μάλλον είναι χρήσιμο να πάρω το λόγο. Θα τα πω στα γρήγορα αλλά ανοιχτά. Για τη δική μου πολιτική ομάδα, ο φάκελος αυτός για την ε, διαλειτουργικότητα είναι και πολιτική προτεραιότητα και τεχνική επιταγή. Και δεν θα πρέπει να στηριχθείτε στη δική μου ομάδα για να αφαιρέσετε το ουσιαστικό κομμάτι από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή για να ακολουθήσετε κάποιες τακτικές κολυσιεργίας για ένα θέμα το οποίο για μας είναι ζωτική σημασίας και θα πρέπει να εγκριθεί πριν το τέλος της δικής μας θητείας. Θεωρούμε λοιπόν πως η πρόταση που πρέπει να συζητηθεί και να τροποποιηθεί είναι ουσιαστικό εργαλείο για να έχουμε περισσότερη ασφάλεια στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκής Ένωση για να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα των ακριβών και πολλών εργαλείων που έχουμε στήσει που χάνουν κομμάτι της αποτελεσματικότητάς τους εάν δεν είναι διαλειτουργικά. Θεωρούμε δε πως έφτασε η στιγμή να αποδείξουμε πως είναι δυνατόν να σεβόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα και κυρίως την προστασία των προσωπικών δεδομένων και παράλληλα να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες απαιτήσει ανταλλαγής πληροφοριών. Έγινε μια πρώτη συνάντηση σήμερα το πρωί, θα είμαι πολύ σύντομος πρόεδρε. Οι τροπολογίες μας νομίζω στηρίχτηκαν σε αρκετό βαθμό από, τους, από τον εισηγητή, δεν θα έλεγα από τις ομάδες. Και έχω ακόμα δύο παρατηρήσεις Πρώτον, η ομάδα μου στηρίζει τη χρήση του, κοινού, του κοινού θεματολογίου ταυτότητας μια και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της πρότασης και δεν θα πρέπει να εξαφανιστεί. Είναι το μόνο εργαλείο που επιτρέπει να καταχωρούμε τους εγκληματίες οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων και τους οποίους δεν μπορούμε να τους συνδέσουμε μεταξύ τους γιατί έχουν διαφορετικές ταυτότητες. Θέλω να μου δείξετε πώς θα μπορούσε να γίνει αν δεν έχουμε αυτή την κοινή βάση την οποία επιδιώκουμε. Βεβαίως μπορούμε να περιορίσουμε τη χρήση ε, αυτής της βάσης από τη στιγμή που θα είναι διαθέσιμη για να μην χρησιμοποιείται υπό οποιασδήποτε συνθήκες από τους ε, ε, αστυνομικού, για παράδειγμα τη στιγμή που προχωρούν σε κάποια σύλληψη ή ε, σε περίπτωση που πρόκειται για ανήλικο που συλλαμβάνεται. Δεύτερον, στα τεχνικά ε, που έχουμε καταθέσει θέλω να μου πείτε είναι σωστό να προσθέσουμε και άλλα δεδομένα πέραν αυτών που έχει η πρόταση της Κομισιόν. Για παράδειγμα, στοιχεία από τη Europol Είμαστε λοιπόν υπέρ του εργαλείου αυτού και αυτό που θα παρακολουθήσουμε είναι να σεβαστούμε όσο γίνεται τις απαιτήσει οι οποίες έχουν επισημοποιηθεί το τελευταίο διάστημα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και λυπάμαι που έκανα λάθος στη σειρά με την οποία έδωσα το λόγο στις ομάδες. Κορνίλη εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Και υπενθυμίζω, γιατί το συζητάμε το θέμα αυτό. Ποιο ήταν το σημείο αφετηρίας. Ήτανε λοιπόν ότι οι εγκληματίες θα πρέπει να εντοπίζονται και να συλλαμβάνονται σύντομα. Αλλά αν ε, κοιτάξουμε τώρα το αποτέλεσμα και παρακαλώ την Άλντε να το σκεφτεί πάλι. Δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται κυρίως έχει να κάνει με πολίτες τρίτων χωρών. Τους οποίους αντιμετωπίζουμε με δυσπιστία δηλαδή. Γιατί αν δείτε τι συμπροματικές βάσεις στοιχείων θα δημιουργήσουμε, τότε διαπιστώνουμε ότι αφορά τους πάντες. Όχι μόνο συγκεκριμένα άτομα. Υπενθυμίζω ότι ο υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων ε, λέει ότι αν τα εφαρμόσουμε όλα αυτά, τότε δεν υπάρχει πλέον δρόμος επιστροφής. Θα δημιουργήσουμε τεράστιες βάσεις δεδομένων που θα λειτουργούν για πάντα. Και θα πρέπει να δούμε αν αυτό επιτυχάνει τη σωστή ισορροπία με την προστασία των ε, θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων. Είχαμε πει ότι θέλουμε να απλουστευτούν οι βάσεις στοιχείων για να επιτύχουν ακριβώς το στόχο τους καλύτερα. Αλλά αυτό που προέκυψε είναι εντελώ διαφορετικό. Και η συζήτηση για τη λεγόμενη απάτη ε, όσον αφορά την ταυτότητα. Είναι λίγα άτομα. Και ακούσαμε από διάφορες ε, ακροάσεις ότι το θέμα αυτό δεν είναι τόσο απλό. Η απάτη ταυτότητας. Ακούσαμε πολλά στοιχεία. Και ξέρουμε ότι πολλά θέματα παραμένουν ανοιχτά και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα είπαμε ότι μειώνεται η ανάγκη απόδειξης σκοπιμότητας, μειώνεται η αυστηρότητα για την πρόσβαση. Θα είχαμε συζητήσει αυτά σχέση με την Interpol και πάλι ξαναπροκύπτουν. Μεγάλο θέμα λοιπόν αυτό. Οπότε νομίζω ότι ο εισηγητής δεν θα θεωρήσει ότι είμαστε επικοδομητικοί γιατί μία πρότασή μας είναι να επιστραφεί αυτή η πρόταση στην Επιτροπή γιατί δεν θεωρούμε ότι εξυπηρετεί το στόχο για τον οποίο ξεκινήσαμε. Λοιπόν, ας πούμε ότι δεν επιστραφεί το θέμα αυτό. Τότε έχουμε άλλες προτάσεις που πιστεύουμε ότι μπορούν να συζητηθούν επικοδομητικά. Και κάναμε πρόταση. Και είπαμε, ωραία, καταλαβαίνω ναι, μπορούμε να φτιάξουμε μια δικτυακή πύλη. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι σωστή η διαλειτουργικότητα. Εάν βελτιωθούν οι κανόνες για την πρόσβαση και για την ε, σκοπιμότητα κάθε έρευνας, μπορεί να βοηθήσουν όλα αυτά. Και αυτό το δεύτερο σημείο, την κοινή υπηρεσία για την, ε, το BMS, για τα βιομετρικά. Και αυτό το καταλαβαίνουμε. Σίγουρα βοηθάει. Βεβαίως θέλουμε να είναι αποκεντρωμένο. Όχι να είναι μία μεγάλη βάση δεδομένων. Μέχρι, εκείς, μέχρι εκεί θα μπορούσαμε να συζητήσουμε συμβιβασμούς. Αλλά αυτό που προκύπτει μετά είναι απόλυτα απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε τις επόμενες βάσεις δεδομένων. Γιατί όλα αυτά είναι απόλυτα δυσανάλογα ο καθορισμός ταυτότητας. Αν διαβάζω αυτά που λέει, τα δεδομένα που λέει αυτό για την ταυτότητα, τι στοιχεία θέλετε να συμπεριλάβετε εδώ μέσα και πώς θα συνδυαστούν. Όλα αυτά τα θεωρούμε ότι είναι απόλυτα απαράδεκτα. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι χρειάζονται. Και για αυτόν τον ε, υπερανιχνευτή των ε, ε, τόσο το, το, τόσο πολλών στοιχείων αυτό θα μας δώσει πολλά αποτελέσματα, πολλαπλά αποτελέσματα. Οπότε στην ουσία θα έχουμε λανθασμένους συναγερμούς. Άρα δεν θα πιάνουμε τους εγκληματίες. Όπως έχει τώρα αυτή η πρόταση, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε μαζί της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Κορνήλια. Λυπάμαι που χρειάστηκε να σε διακόψω. Έχουμε ακόμα τρεις κοιόδεις. Φραντς Βελέρο και Βίκστρομ. Μπορείτε να με βοηθήσετε, συνάδελφοι. Μπορείτε να περιοριστείτε στα δύο λεπτά, κυρία Στίβεν? Επίσης και κυρία Στίβεν, από δύο λεπτά, για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στις 6. Ξέρω πως μπορείτε να πείτε πολύ περισσότερα για το θέμα αυτό, αλλά σήμερα παρακαλώ περιοριστείτε για... Στα δύο λεπτά, ο κύριος Φράντ για τους πράσινους. Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα αυτό μπορεί να φαίνεται πολύ τεχνικό, αλλά είναι ιδιαίτερος πολιτικό. Η Επιτροπή προτείνει όλες οι βάσεις δεδομένων για τη διαχείριση της αστυνομίας και των συνόρων, να τις συνδυάσουμε και να έχουμε ένα, και ένα κεντρικό μητρό για την ταυτότητα. Όπως σωστά λέει ο υπεύθυνο για τα προσωπικά δεδομένα. Αν κάνουμε κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει πλέον επιστροφή. Αυτή, αυτές οι βάσεις έχουν δημιουργηθεί για ε, διαφορετικούς σκοπούς. Πρέπει λοιπόν να μείνουν χωρισμένες. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της οι υπεύθυνοι για τα σύνορα πρέπει να κάνουν τη δική τους και οι υπεύθυνοι για τη μετανάστευση τη δική τους. Γιατί για κάθε βάση δεδομένων πρέπει να υπάρχει ε, η αναγκαία απόδειξη της ανάγκης για τη χρήση της. Η γερμανική ταυτότητα, για παράδειγμα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και επιγραμμικά, έχει διάφορα ψευδόνυμα ανάλογα με τον λόγο χρήσης αυτό το κοινό ε, μητρό ταυτότητας θα τα καταργήσει όλα αυτά. Η Κομισιόν δεν απέδειξε μέχρι τώρα την ε, αναγκαιότητα και την αναλογικότητα όλης αυτής της σύνδεσης. Σας παρακαλώ, αναφερθήκατε στον Άννη Σάμρη που έκανε αυτή την επίθεση στο Βερολίνο και είχε 14 διαφορετικές ταυτότητες. Ήταν γνωστός από τις αρχές και τον παρακολουθούσαν. Και αυτό που πήγε στραβά στην προσπάθεια των αρχών το εξετάζει μία επιτροπή ε, της ε, Γερμανικής Βουλής. Και σίγουρα δεν ήταν το πρόβλημα, δεν το γνωρίζαμε. Οι διάφορες τράπεζες δεδομένων, τα συστήματα αιτιάς και εισόδου-εξόδου δεν χρειάζονται να έχουν ε, δεν θα χρειάζονται τότε αλλά θα βασίζονταν σε ένα κεντρικό δεδομένο ένα κεντρικό, μια κεντρική βάση γι' αυτό θέλουμε αυτό το κεντρικό σύστημα να καταργηθεί όπως το ζητάνε και οι σοσιαλιστές και οι γκουε αυτό που θα μπορούσαμε να δεχθούμε θα ήταν αυτό, αυτή η ενιαία δικτυακή πύλη για τις ε, αναζητήσεις, αλλά αυτό είναι ήδη ε, μεγάλη παραχώρηση από, τις, ε, από πλευράς μας, γιατί όπως ξέρετε για βασικούς λόγους μας τα κατά διαφόρων βάσεων δεδομένων. Δεν χρειάζομαι δύο λεπτά. Συμφωνώ με αυτά που είπα προηγούμενο. Ευχαριστώ πολύ, Μποντίν. Η Σεσίλια για την Άλντε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Κλοντ. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω όλους. Ελπίζω να περάσετε καλά το καλοκαίρι, γιατί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των ε, συστημάτων δεδομένων αποτελεί ένα σημαντικό ε, στοιχείο στο οποίο δεν έχουμε εκμεταλλευτεί στο έπακρο και γι' αυτό είναι σημαντικό να προχωρήσουμε. Πιστεύω και πάντα πίστευα στην ανταλλαγή πληροφοριών και μαζί με την πολιτική μου ομάδα πολύ συχνά έχουμε πει πως θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική. Η διαλειτουργικότητα όμως δημιουργεί και τεχνικά και πολιτικά θέματα και προκλήσεις. Σίγουρα θα καταφέρουμε να τα ξεπεράσουμε, όμως μπορεί να χρειαστούμε χρόνο. Επίσης, γιατί κάποια από τα συστήματα τα οποία θα συμπεριληφθούν αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό αναθεώρηση και αυτό δημιουργεί και πιο συγκεκριμένα προβλήματα. Οι προτάσεις αυτές προσθέτουν άλλο ένα στρώμα ε, επιπλοκών σε θέματα τα οποία ήδη είναι περίπλοκα. Ο στόχος είναι να σεβαστούμε ε, την αναλογικότητα, την αναγκαιότητα και παρόλα αυτά να προχωρήσουμε. Οι τροπολογίες οποίες έχω καταθέσει σκοπεύουν στο να βελτιώσουν το κομμάτι των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την προστασία των δεδομένων, όπως επίσης και την ενημέρωση των ατόμων των οποίων αποθηκεύονται τα δεδομένα. Και στα πλαίσια αυτά θεωρώ πως είναι σημαντικό εμείς να ακούσουμε τις υπηρεσίες μας όλες τις σχετικές με τα θέματα αυτά και να συμπεριλάβουμε και κάποιες διατάξεις την προστασία των παιδιών αλλά και των υπηκών τρίτων χωρών. Θεωρώ επίσης σημαντικό να έχουμε και κάποιες δικλείδες ασφαλείας έτσι ώστε να μην γίνονται παραβιάσεις και κυρίως για τα όσα αποκαλύφθηκαν στην αξιολόγηση τη χρήση του συστήματος έγκαινα από διάφορα κράτη-μέλη. Ασφαλείς λοιπόν ρυθμίσεις έτσι ώστε κάθε κράτος μέλος να συμμορφώνεται απόλυτα με τους κανόνες που έχουν περιγραφεί για κάθε ένα από τα συστήματα τα οποία θα αποτελέσουν κομμάτι ε, της διαλειτουργικότητας. Με χαρά περιμένω την εκκίνηση των διαπραγματεύσεων για να καταλήξουμε στον καλύτερο δυνατόν συμβιβασμό και να σεβαστούμε τα δικαιώματα των πολιτών μας στην ιδιωτική του ζωή, εξασφαλίζοντας όμως ασφάλεια για όλους. Αυτό γίνεται και γι' αυτό περιμένω να δω ε, τα πόσα θα πετύχουμε ε, στις προσπαθίες μας. Ευχαριστώ πολύ Σεσίλια. Να προτείνω... Α, συγγνώμη, κυρία Στίβενς. Ε, θα εκπροσπίσω τον κύριο Ντάλτον αν δεν κάνω λάθος. Και νομίζω είστε και η τελευταία. Είμαι, ο αντικαταστά... Είμαι η αντικαταστράτρια του κύριου Ντάλτον και έχω να σας πω πως Έχουμε θέματα ασφάλειας, θέματα διαχείρισης συνόρων και γι' αυτό χρειαζόμαστε πιο ευφυή χρήση των πληροφοριών που είναι ήδη διαθέσιμες από τις αρμόδιες αρχές. Η διαλειτουργικότητα θα πρέπει να προσφέρει μία ε, επιπρόσθετη αξία και να είναι αποτελεσματική, αποδοτική και ασφαλής. Ανησυχώ πάντως για τις τροπολογίες που έχουν υποβάλει ε, κάποιες ε, πολιτικές ομάδες που θέλουν να διαγράψουν το CIR που είναι η κοινή βάση. Γιατί αν κάνουμε κάτι τέτοιο το όλο σύστημα θα γίνει λιγότερο αποτελεσματικό, θα γίνει πιο περίπλοκο και θα έχει και περισσότερο κόστος. Δηλαδή, επιπλέον βάρος για το σύστημα και για τις αρχές που χρησιμοποιούν τα συστήματα αυτά. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το να έχουμε αυτή τη νέα κοινή βάση, δεν σημαίνει πώ θα κατέψουμε όλα τα δεδομένα. Όχι. Θα έχουμε μία πλατφόρμα στην οποία τα δεδομένα από τι διάφορε βάσει ε, θα συμπεριλαμβάνονται με σαφέστατε διακρίσει πρόσβαση και προστασία. Ευχαριστώ που ήσασταν τόσο σύντομοι. Ξέρω πως οι συγητές μας άκουσαν τα σχετικά ε, σημεία. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να αποβαντήσετε γιατί έχουμε και τις ψηφοφορίες. Πάντως θέλω να λάβετε υπόψη τα όσα ακούσατε. Ξέρω πως μέχρι τις 10 Οκτωβρίου θα γίνει μια σειρά συναντήσεων. Οπότε ξέρω πως ακούσατε και τα όσα σας είπαν οι Μέχρι λοιπόν τις 10 του μηνός ελπίζω, σας εύχομαι μάλλον καλή τύχη γιατί ξέρω πως είναι πολλές οι τροπολογίες και σας ευχαριστώ για το έχετε κάνει μέχρι σήμερα. Κύριε Λέναρς, κύριε Μέλος, σας ευχαριστώ. Και περιμένω και τα αποτελέσματα. Ωραία λοιπόν. Και ευχαριστώ και τους σκιώδες βέβαια. Τώρα λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Καθίστε, ετοιμαστείτε και θα προχωρήσουμε στην πρώτη ψηφοφορία. Κυρία Κάφμαν. Λοιπόν, εδώ που κάθεστε θα σας υπενθυμίσω πως στην τρίτη ψηφοφορία που θα κάνουμε θα πρέπει να πάμε σε άλλη αίθουσα γιατί ψηφίζουμε μαζί με την ΕΚΟΝ. Και βέβαια μην ξεχάσετε τις κάρτες σας. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Περνάμε στην ψηφοφορία. Λοιπόν, συνάδελφοι, να περάσουμε στην πληροφορία, Η Αντιπρόεδρε, κυρία Γκουτζίσκα, θέλει να κάνει μια πολύ σύντομη παρέμβαση. Μπάρμπαρα, παρακαλώ. Αύριο στις 6.30 έχουμε αυτή την έκθεση για την αγώνα των Πολωνών για τη δημοκρατία. Σας παρακαλώ να έρθετε στην έκθεση και τη συζήτηση. Θα γίνει συζήτηση μετά. Είναι πολύ σημαντικό να φανεί, να φανεί ότι ενδιαφέρεστε για τους Πολωνούς. Είναι πολύ σημαντικό για τους Πολωνούς που συμμετέχουν στις ε, απεργίες και διαδηλώσεις. Παρακαλώ ελάτε στην ε, έκθεση και τη σύντομη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ Μπάρβαρα κύριε Λόπεθ Αγγιλάρ. Περιμένω εδώ και 10 λεπτά να μου φέρουν την ηλεκτρονική μου ε, κάρτα ψηφοφορίας. Α, νόμιζα πως θα τα κάτι το συναρπαστικό, αλλά τελικά όχι. Ωραία, λοιπόν. Περνάμε στη ψηφοφορία. Συμβαστική σχέδιο έκθεσης για την καταπολέμηση της απάτης και της παραχάραξης μη ε, ε, πληρωμών με μη, όχι με χαρτονομίσματα και νομίσματα. Η κυρία Κάφμαν, ευχαριστώ τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν και τους βοηθούς και τους συναδέλφους όλους και τη γραμματεία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συμβαστική C, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 1. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική για το άρθρο 3. Άρχεται. Πέρα. Δεκτή. Συμβαστική για το άρθρο 4. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική για το άρθρο 5. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 101. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 16. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 102. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 103 Όχι 103. Ωραία, πάμε λοιπόν στο, στη συμβαστική για το άρθρο 7. Όχι, 103. Λοιπόν, πάμε στην ε, συμβαστική επί του άρθρου 7. Άρχεται. Πέρα. Δεκτή. Συμβαστική για το άρθρο 8. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική για το άρθρο 10. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική για το άρθρο 11. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική για το άρθρο 12. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική για το άρθρο 13. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική για το άρθρο 14, το άρθρο 16α και το 23α. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική για το άρθρο 15 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική για το άρθρο 16. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 170. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 171. Άρχεται. πέρας δεκτή 173 άρχεται πέρας δεκτή συμβαστική για το άρθρο 19 άρχεται πέρας δεκτή συμβαστική για το άρθρο 20 άρχεται πέρας δεκτή. Αιτιολογικές σκέψεις, τροπολογία 30, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική α, άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική β, άρχεται. Πέρας δεκτή. Τροπολογία 35 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 36 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 38 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 39. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική D. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική ε. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική F. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική G. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική Ήτα. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 57. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική γιώτα άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική J άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική K άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική L άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική μη. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική νη. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία εννέα, Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική όμικρον. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική ρο. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική Q. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 74. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική, ε, συγγνώμη, τροπολογία 75 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τελική ονομαστική άρχεται. Πέρας. Δεκτή 31 ψήφοι υπέρ, 1 κατά, 0 αποχές. Και η τελική ψηφοφορία για απόλυτη πλειοψηφία με βάση τον κανόνα 69 άρχεται. Άρχεται λέγω. Χρειαζόμαστε 31 ψηφοφορίες. Συνεχίζεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. 31 ψήφους χρειαζόμαστε. 37. Ωραία. Και μία ψήφος κατά. Ωραία. Συγχαρητήρια. Την κυρία Κάφμαν. Να περάσουμε στην επόμενη έκθεση. Κατευθείαν η κυρία Φεράρα είναι η συγγήτρια. Είναι η απόφαση σχετικά με τη σύναψη από την Eurojust Συμφωνία για τη συνεργασία μεταξύ της Ιδίας και της Αλβανίας. Θέλετε να πάρετε το λόγο πριν την ψηφοφορία, όχι. Να προχωρήσουμε λοιπόν αμέσως, δεν υπάρχουν τροπολογίες, πάμε στην τελική ψηφοφορία που θα πρέπει να γίνει με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 34 ψήφους υπέρ, μία κατά και τρεις αποχές. Συγχαρητήρια στην κυρία Φεράρα. Uh, uh, Συνάδελφοι, να ανακοινώσω μόνο ότι τώρα όσοι θα ψηφίσετε θα πάμε στην Επιτροπή, ε, στην Επιτροπή PHS 3C50, στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Αν πάμε γρήγορα, μπορούμε να τελειώσουμε σύντομα. Γρήγορα όλοι λοιπόν στην 3C50.